Yeah, so what did you What did you working what came to see the... Buonasera a tutti. Καλησπέρα σας, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να αρχίσουμε με τα συνηθισμένα. Τότε δηλαδή θα μεταδοθεί η συνεδρίαση στο διαδίκτυο. Το πρώτο σημείο μας είναι η έγκριση της μίλησας διάταξης που σας έχει διανεμηθεί στις 6 Δευτέρου του 2013. Και σας υπενθυμίζω ότι ξεκινήσαμε καθυστερημένα λόγω του ότι έπρεπε να αρχίσουμε στις 3.30 μια, μια που είχαμε τη συνεδρίαση των ε, Προέδρων, στη διάσκεψη των Προέδρων. Πήγα εγώ τελείωσε στις 3.30. Τέλος πάντων, ξεκινούμε τώρα και προχωρούμε. Οι τροπολογίες για την έκθεση για να πάρα παραπολές και η συζήτηση είναι περίπλοκη όσον αφορά τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα οπότε δεν μπορούμε να κάνουμε την ε, ε, ψήφιση στις 19 Φεβρουαρίου αύριο όπως είχαμε πει οπότε θα δούμε σήμερα όταν τελειώσει η συζήτηση ποια θα είναι η ημερομηνία για να γίνει αυτή η ψηφοφορία. Ετήση του κυρίου Σέφλιν και του κυρίου Νταφ όσον αφορά την έκθεση για την ε, τσεχική δημοκρατία. Αυτό θα συζητηθεί με άλλη σειρά από ό,τι είχαμε πει για σήμερα. Τώρα όσον αφορά την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση έχουμε την έκθεση αυτή η οποία ε, θα αναπαιμφθεί. Οπότε, θα αλλάξει και αύριο κάπως οι ε, συνεδρίαση στις 9 θα αρχίσουν, θα αρχίσουν η συζήτηση και τελειώσουν στις 3 και θα τελειώσουν οι συνεδρίασεις 9 με 10 και μισή και μετά πάμε μέχρι τις 3. Οπότε, έχουμε τώρα την έκθεση για την Τσεχική Δημοκρατία και για την πολιτική κυβέρνηση, δεν μπορούμε να το συζητήσουμε. Και δεύτερο σημείο, η ανακοίνωση του Προέδρου, δεν έχω και πολλά να σας πω. Σας ενημερώνω απλώ ότι στη συνεδρία της 7ης Δευτέρου οι συντονιστές συμφώνησαν σύμφωνα με την πρόταση της διάσκεψης των Προέδρων, το να γίνει αυτή η έκθεση δύο πρωτοβουλίας όσον αφορά την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και δέχθηκαν το έτοιμά μας να έχουμε δύο συνεισηγητές. Το ECR και η Πράσινη το ανέλαβαν και θα είναι αυτοί οι κύριοι Φόξ και Χέφνερ. Στις 26 Φεβρουαρίου σας θυμίζω προβλέπεται να γίνει έκτακτη συνεδρίαση και πρόκειται επίσης να έχουμε αυτήν την ε, διάσκεψη για το παρατηρητήριο που είναι δραστηριότητα του κέντρου Ρόμπερτ Σούμαν του Πανεπιστημιακού Ευρωπαϊκού Ιδρύματος. Πρώτα απ' για τα πολιτικά ιδρύματα και το δεύτερο όσον αφορά τα εκλογικά δικαιώματα των Ευρωπαίων. στι 26 Οκτωβρίου θα γίνει αυτή η τη συνεδρία. Και τώρα, όσον αφορά τα πρακτικά, σας έχουν ε, διανεμηθεί για 26-27 Νοεμβρίου. Εάν δεν έχετε κάποιες παρατηρήσεις, εγκρίνονται. Οπότε και τώρα προχωρούμε στο κυρίως θέμα μας. Αυτό που το είχαμε στους ανέξει και είναι αυτό το σχέδιο πρωτοκόλλου για την εφαρμογή του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Τσεχική Δημοκρατία. Οπότε θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Νταφ. Έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα σε όλους πρώτα-πρώτα και σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε για πολλωστή φορά να μιλήσουμε για αυτό το πρωτόκολλο. Το πρωτόκολλο το οποίο θα προσαρτηθεί στον χάρτη των δικαιωμάτων. ό,τι γνωρίζω, σύμφωνα όλες οι πολιτικές ομάδες. Ούτως τώρα για τρίτη φορά να προβούμε σε ψηφορία. Έχουμε δύο, τρεις μάλλον, σημαντικές αλλαγές στην έκθεση. πρώτα-πρώτα στην αιτιολογική έκθεση, στην αυτή παράγραφο. Επισημαίνεται στο Συμβούλιο, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ότι δηλαδή θα πρέπει να συνενέσουν στην τροποποίηση της συνθήκης παρά τις προδοποιήσεις, τις επιφυλάξεις, ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ότι δηλαδή το σωστό θα ήταν τα άλλα κρατημέλη να μην αρχίσουν τη διαδικασία της κύρωσης πριν γίνει αυτή η διαδικασία από την Άνω και Κατοβουλή στην Τσεχία και πριν ολοκληρωθεί εκεί. Και ο λόγος προς τούτο είναι ότι σαφώς είναι πάρα πολύ αβέβαιο το ότι θα δημορφωθεί η κατάλληλη πλειοψηφία στην Πράγα. Ούτως ώστε να ολοκληρωθεί η κύρωση ή τέλο πάντων η τροποποίηση της συνθήκης σε σχέση με αυτή την παρέκκληση που αφορά την ε, εφαρμογή του χάρτη από τα τσεχικά δικαστήρια, όπως γνωρίζετε. Η κατάσταση εκεί μεταβάλλεται. και υπό τη νέα σύνθεση στην Άννα και Καταβούλια ίσως τα πράγματα πάρουν κάποια απρόβλητη τροπή. Η δεύτερη μεταβολή τώρα αφορά την πρώτη παράγραφο. Δεν να πούμε συμφωνούμε ή δεν συμφωνούμε την πρόταση, απλώς λέμε ότι αναγνωρίζουμε, διαπιστώνουμε τη διαβούλευση με το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τις συνθήκες. Τέτοια αλλαγή υπάρχει στην δεύτερη παράγραφο εκεί όπου λαμβάνει την εντολή ο πρόεδρος να προωθήσει το ψήφισμά μας που αποτελεί τη θέση του Κοινοβουλίου να το προωθήσει λίγο προς το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Πρόκειται επίσης για κάποια πιο ουδέτερη διατύπωση, οπότε και εμείς ως Επιτροπή μπορούμε να εγκρίνουμε το κείμενο με μια ισχυρή πλειοψηφία αύριο. Και να μην απονευρώνουμε το κείμενο, ούτε να αποδυναμώνουμε τη, την επιχειρηματολογία του κειμένου ή των αιτιολογικών παραγράφων. Και τι επομένως μπορούμε να κατέβουμε έτσι με το κείμενο αυτό στην ε, Ολομέλεια του Μαρτίου και έτσι να ολοκληρωθεί η διαδικασία μαζί. Για αυτό το κείμενο και όπως είδατε στην λίστα της ψηφοφορίας έχω λάβει υπόψη τις ε, τροπολογίες του ECR αφού τις μελέτησα με μεγάλη προσοχή και αυτό που προτείνω είναι να καταψηφιστούν. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Ποιος θέλει το λόγο. Έχετε το λόγο, κύριε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Τρίτη φορά είναι που το συζητάμε αυτό το ε, τσεχικό πρωτόκολλο. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Δάφ, έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Τον ευχαριστούμε γι' αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην ίδια παράγραφο, στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο εισηγητής, όσον αφορά τη διαδικασία κύρωσης. Ε, προτείνεται να ε, ξεκινήσει κάτι τέτοιο στην Τσεχία για πρακτικούς λόγους η τσεχική γερουσία εδώ και πολύ καιρό ήταν απρόθυμη ε, για την έγκριση τη εξαίρεση του πρωτοκόλλου αυτού για τα ανθρώπινα τα δικαιώματα, γιατί θεωρεί ότι μπορεί αυτό να θέτει την αμφιβόλο τα δικαιώματα των ε, τσέχων πολιτών και θεωρεί ότι τότε οι ε, πολίτες δεν θα είχαν τα ίδια δικαιώματα με τους πολίτες άλλων χωρών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα προτείνω να καταψηφίσουμε αυτήν ε, την ε, τροπολογία, πρέπει να αρχίσει η διαδικασία κύρωσης ε, στην τσεχική δημοκρατία. Νομίζω ότι όπως έχει τώρα η έκθεση πρέπει να την υποστηρίξουμε. Δεν τάσσομαι υπέρ της πλήρους απόρριψής Thank you, Ευχαριστώ πολύ. Μας είπε ο κύριος Δαφ ότι είναι η νιωστή φορά, η νιωστή φορά στο τετράγωνο να μην πω εγώ, στον κύβο. Είναι πολλωστή φορά τέλο πάντων όσο καιρό είμαι εγώ εδώ που το έχουμε συζητήσει αυτό το πράγμα. Ε, ήταν εξαιρετική η δουλειά του ε, ε, κυρίου Νταφ. Μπορείτε να βάλετε μία Ο κύριος Ντάφ έχει ήδη αναφερθεί ε, στις πολιτικές εξελίξεις στην Τσεχική Δημοκρατία που είναι ε, κατά πολλές έννοιες ε, πολύ σημαντικός παράγοντας. Πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία κύρωσης στην Τσεχία και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα καθυστερήσει βέβαια και η κύρωση. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, αυτά έχει η πολιτική. Αυτά έχω να πω το έχουμε συζητήσει άλλωστε πάρα πολλέ φορέ. Φαίνεται πάντως ότι τελικά τα opt-out δημιουργούν πολλά προβλήματα πάντοτε. Onorevole prego, parola. Chairman, thank you κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα και εγώ να μιλήσω για τις ε, τροπολογίες ε, εξ ονόματος Ashley Fox ε, και άλλων. Κατά τη διάρκεια της συνδίκη Λισαβόνας, οι Βρετανοί ψηφοφόροι είχαν πει, είχαν, τους είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα ίσχυε ο χάρτης μελλοντών δικαιωμάτων για τους Βρετανούς πολίτες δεσμευτικά. και τότε, όταν ζητήσαμε την άποψη του δικαστηρίου, μάθαμε ότι τελικά τελικά η χάρτα και θεμελιωδών βιωμάτων όντως ισχύει ε, στο ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα λοιπόν να καταστήσω σαφές τι σημαίνει κάτι τέτοιο. Όταν μιλάμε για ε, τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όλες ε, οι υποσχέσεις της πολιτικής τάξης πρέπει να θεωρούνται ίσες για όλους. Όμως υπήρξαν πάρα πολλά ψεύδη και μιλάω για την τροπολογία 5. Το γεγονός ότι η Χάρτα και Δικαιωμάτων όντως ισχύει και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όταν μιλάμε για ευρωπαϊκό δίκαιο, το γεγονός ότι είπε ο κύριος ε, Νταφ δεν είναι μία άποψη, είναι γεγονός. Και η ε, κατάργηση της τροπολογίας 5 είναι ουσιαστικά σαν να προσπαθούμε να κρύψουμε κάποια πράγματα από τους ψηφοφόρους ε, στην Πολωνία και στο Ηνωμένο Βασίλειο Κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι λάθος. Ε, έχουμε εκλογές το 2014 και εμείς δεν θα ξεχάσουμε το γεγονός ε, ότι ε, δεν είναι δυνατόν οι ψηφοφόροι να μην γνωρίζουν σοβαρά στοιχεία για αυτό το θέμα. Δεν έχω τελειώσει. Άντριο, αυτό σε αφορά. Μου έκανε πολύ εντύπωση ότι εγκρίνω κάτι το οποίο λέει ο κύριος Νταφ, κάτι το οποίο σπανίω συμβαίνει. είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια των συντηρητικών πολιτικών ε, στη Βρετανία να ε, κρύψουν ορισμένα πράγματα, γιατί για ποιο άλλο λόγο θα ήθελαν να διαγραφεί η τροπολογία 5. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μέσερ Ευχαριστώ. Να απαντήσω σύντομα. Εγώ είμαι από χώρα που έχει εμπειρία στις εξαιρέσεις και μάλιστα τώρα το συζητάμε σε σχέση με το ευρώ την εξαίρεση. Η έκθεση του κυρίου Ντάφ, λοιπόν, δεν βρίσκει το στόχο της, γιατί πρέπει να ξέρουμε το στόχο που είναι η ανησυχία, η μεγάλη μεταξύ πολλών Ευρωπαίων πολιτών που βλέπουν το κράτος πρόνοιας να στοχοποιείται λόγω της εσωτερικής αγοράς, της ελεύθερης διακίνησης εργαζομένων και λόγω αυτού του χάρτη και των κοινωνικών επιπτώσεων. Μπορεί να διαφωνούμε εδώ για το αν αυτό ισχύει και ότι αν στοχοποιείται το κράτος ε, πρόνοιας, αλλά πολλοί πάντως το νιώθουν αυτό, είτε είναι αλήθεια είτε όχι. Αντί να τους παραμερίζουμε και να λέμε ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν δικαιώματα και δεν πρέπει δηλαδή να λαμβάνουμε υπόψη τις ανησυχίες τους, πρέπει να ασχοληθούμε ακόμα περισσότερο γιατί μπορεί και να έχουν κάποιο δίκιο. Η έκθεση του κυρίου Ντάφ κάνει το εντελώς αντίθετο και λέει όποια και αν είναι η ανησυχία στην τεχνική δημοκρατία, όποια είναι η ανησυχία των ψηφοφόρων, κάνουν λάθος. Και γι' αυτό το πρωτόκολλο δεν το επηρεάζει. Δεν επηρεάζει. Από πολιτική άποψη, δεν είναι σοφό αυτό. Πιο σοφό είναι να κάνουμε συζήτηση με αυτούς που ανησυχούν είτε συμφωνούμε είτε όχι μαζί τους. Αλλά και από νομική άποψη νομίζω ότι είναι λάθος προσέγγιση, γιατί σε τελευταία ανάλυση δεν θα είναι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα κρίνει και θα αξιολογήσει το περιεχόμενο του πρωτοκόλλου αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε πολλές ε, περιπτώσεις ε, νομικές υποθέσεις στο Λουξεμβούργο που εξετάζονται για το περιεχόμενο κάποιων πρωτοκόλλων που μπορούν να συμφωνηθούν ε, με τη διαδικασία. Και αυτό θα γίνει και εδώ, αν υπάρξει αμφισβήτηση. Ε, στα σημεία LKM, εκεί το Κοινοβούλιο ε, μπορεί να αποφασίσει ότι το πρωτοκόκολο ανεξάρτητα από την απόφαση του δικαστηρίου δεν θα έχει αποτέλεσμα κλπ. Εδώ νομίζω ότι από νομικής άποψης είναι κακή πρακτική ένας τέτοιος ε, ισχυρισμός. Εγώ θα ταχθώ υπέρ των τροπολογιών ECR και αν απορριφθούν θα πρέπει, λυπάμαι που το λέω Άντριου, να καταψηφίσω και όλη την εκθεσή σου. Ευχαριστώ. Άλλες. Ο συνάδελφος Έφνερ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κάποιες ιστορίες δεν τελειώνουν ποτέ. Έχει δίκιο ο συνάδελφος Σέφλιν. Υπάρχουν όμως και άλλες ιστορίες που δεν θα έπρεπε ίσως να αρχίσουν καν. Και μου φαίνεται ότι αυτό ισχύει με την περίφημη τσεχική εξαίρεση opt-out γιατί νομικά και ουσιαστικά δεν έχει νόημα. Ενώ μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές αμφιβολίες στον πληθυσμό και στη νομική πρακτική και θεωρία σχετικά με το πρωτογενές δίκαιο, τις ευρωπαϊκές συνθήκες, δημιουργώντας ε, αυθαιρεσίες χωρίς να, χωρίς να διασφαλίζει αυτό που ήθελε τότε ο Τσέχος πρόεδρος και που είχε υποσχεθεί ως συνέπεια του opt-out της εξαίρεσης. Δεν υπήρχε ε, στήριγμα στην πραγματικότητα, γι' αυτό ήταν μια ψευδοπολιτική αυτή η πολιτική της εξαίρεσης και δεν πρέπει να συμμετέχουμε σε τέτοιες πρακτικές νομίζω. Εγώ ε, προσυπογράφω τους επένους προς τον εισηγητή τον κύριο Ντάφ, ο οποίος και με τρόπο ευφυή και επίμονο για το Κοινοβούλιο, πιστεύω, προχωρεί το ζήτημα αυτό. Πιστεύω ότι είναι σημαντικό στη γνωμοδότησή μας να πούμε καθαρά ότι ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης, πριν από την έναρξη της διαδικασίας κύρωσης στα κράτη-μέλη, πρέπει να περιμένουμε και να δούμε η... Τα δύο νομοθετικά σώματα του... της Τσεχικής Βουλής θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι θα κάνουν. Ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες εκλογές, νομίζω ότι περισσότερο και από πριν πρέπει να θέσουμε το ερώτημα πώς θα αξιολογήσουμε από νομική άποψη το θέμα ότι εδώ ε, διαπραγματευόμαστε μία επιφύλαξη η οποία δεν διατυπώθηκε από τον τσεχικό λαό ε, δεν ε, παρουσιάστηκε ως επιφύλαξη του τσεχικού λαού, αλλά το τότε πρόεδρος ε, ο Τσέχος Κλάους ε, σε μια μετέπειτα, ε, σε, μια όψιμη διαδικα... σε ένα όψιμο στάδιο της διαδικασίας έθεσε το θέμα, μετά άλλαξαν πολλά, άλλαξε και στο κοινοβούλιο και στην πολιτική της Τσεχίας άλλαξαν πολλά. Άρα νομίζω ότι επιβάλλεται να δούμε πρώτα ποια είναι η πραγματική επιθυμία του τσεχικού λαού και το λέω αυτό κυρίως προς τον συνάδελφο Μέσερ Σμιτ που δεν θέλει να παραγνωρίσει τις ανησυχίες και τις επιθυμίες του τσεχικού λαού, ακριβώς επειδή θέλουμε να τις λάβουμε υπόψη μας, θέλουμε να ξέρουμε ακριβώς τι σκέφτονται οι άνθρωποι εκεί. Και πριν αρχίσουν άλλα κράτη-μέλη τη διαδικασία κύρωσης, να προχωρήσει η Τσεχία. Ε, ε, εγώ συμφωνώ με το σχέδιο έκθεσης Έχω μιλήσει πολλές φορές και έχω εκφράσει τη γνώμη μου σε προηγούμενες φάσεις της διαδικασίας, οπότε ε, εδώ μπορώ να είμαι σύντομος. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Μπρόντς. Το πρωτόκολλο 30 δεν είναι opt-out είπαμε, αλλά τι είναι το δικαστήριο είπε ότι δεν είναι opt-out γενική εξαίρεση και η γενική εισαγγελέα, όχι όμως το δικαστήριο το αυτό. Το δικαστήριο έδωσε μια εξήγηση. Αν είναι εξήγηση, τότε γιατί υπάρχει τόση μεγάλη αντίδραση σε αυτήν. Φαίνεται ότι οποιαδήποτε ψήφος θα αφορά την εφαρμογή ενός πράγματος του οποίου τη φύση δεν καλό καταλαβαίνουμε. Αν το πρωτόκολλο 30 δεν είναι γενική εξαίρεση opt-out, τότε τι σκοπό είχε ε, αυτοί που το σχεδίασαν κάτι ήθελαν να το κάνουν. Αλλά φαίνεται ότι οι συντάκτες του πρωτοκόλλου ήξεραν πολύ καλά ότι δεν είχε καμιά αξία και σκοπό είχε να παραπλανήσει <clears throat> το εκλογικό σώμα κυρίως στην Πολωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο και μετά και στην Τσεχία. Αν ισχύει αυτό, δεν πρέπει απλώς να το κρύψουμε ή να το αντιμετωπίσουμε το θέμα σαν να είναι ίσον. Ε, μπορεί, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι η θελημένη παραπλάνηση της κοινή γνώμης από τον τότε Πρωθυπουργό. Και αυτό βεβαίως έχει τεράστια σημασία και είναι κάτι το οποίο πρέπει να μην διαφύγει της δικής μας προσοχής και της προσοχής άλλων. Δεν θα μπω στη συζήτηση στο εσωτερικό της Τσεχικής Δημοκρατίας, δική τους υπόθεση είναι αυτή, αλλά δεν νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να τους στερήσουμε το δικαίωμα επιλογής που θα έπρεπε ελευθέρως να μπορούν να κάνουν. Ευχαριστώ. Τελείωσαν οι παρεμβάσεις όλες, οπότε ο κύριος Ντάφ τώρα, αν θέλει να δευτερολογήσει. Σας ευχαριστώ και εγώ έχω εκπλαγεί. με το ότι οι Βρετανοί συντηρητικοί θέλουν να τοποθετηθούν υπέρ αυτών των κόλπων που έκανε επί των ημερών του ο κύριος Μπλερ σε σχέση με την αυτοεξαίρεση της Βρετανίας. Μα θεώρησε ότι το σωστό είναι να αναθεωρήσουν την τροπολογία τους. Για τον κύριο Μέσα Σμιτ έχω να πω ότι συμφωνώ. Ότι θα πρέπει να γίνει μια ζήμωση, μια συζήτηση και έχω απευθυνθεί σε πολλούς εκπροσώπους της κοινωνίας, νομικούς, υπουργούς από την χώρα αυτή διπλωμάτες και από τις δύο βουλές. Και με κυβέρνηση και με αντιπολίτευση. Και με εκπροσώπους του συνταγματικού δικαστηρίου του Μπρινού. ουδείς δε από εκείνους είπε Αποστηρίστε μου. Τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τον χάρτη θύμιλο των δικαιωμάτων. Κανείς δεν είπε. Ας έχουν διαφορετική μεταχείριση από τους υπολείπους Ευρωπαίους. Οπότε με αυτά τα δεδομένα πιστεύω ότι η προσέγγιση μας είναι δίκαιη, ε, ενδελεχής. Και στα δύσκολα της πολιτικής, ξέρετε, έχω κολυμπήσει στα βαθιά νερά πολύ καιρό. Παρ' όλα αυτά όμως, τα σε επιμελίας των Πανεπιστημιακού δεν τα έχω ξεχάσει. Πολύ ωραία και έτσι ολοκληρώνεται η συζήτηση για αυτό το θέμα, για το οποίο πρέπει αύριο το πρωί να γίνει η ψήφιση. Και τώρα, προχωρούμε τώρα. το θα είμαι σήμερα στη διατάξη, έχουμε τώρα την έκθεση της κυρίας Γιαννάκου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, το σημείο, το σημείο 4. το έχουμε συζητήσει για μικρό να έχουμε τις τροπολογίες. Οπότε και μπορούμε τώρα να δούμε εις βάθος τι ισχύει για το σημαντικό αυτό θέμα. Εάν θέλει τώρα, ας λάβει το λόγο η κυρία Γιαννάκου. Να ακούσουμε ευχαριστώ για άλλη μια φορά και να σας ευχαριστήσουμε για το έργο το οποίο το έχετε επιτελέσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Όπως ε, είχαμε τονίσει και την τελευταία φορά, υπάρχουν 370 τροπολογίες εκ των οποίων 100 περίπου έχουν ενσωματωθεί σε 20 ε, συμβιβαστικές τροπολογίες τις οποίες χρειάζεται να βούμε με προσοχή και οι άλλες βέβαια εάν περάσουν συμβαστικές πιθανόν να εκπέσουν ή και να ψηφιστούν και αυτές όπως γίνεται συνήθως. Επειδή το λεπτό θέμα της υπόθεσης βρίσκεται Πρώτον, στο, στην καταγραφή του κόμματος, στο registration. Δεύτερον, στον ετήσιο έλεγχο. Και τρίτον, στο τι κάνει το Κοινοβούλιο ή τα ευρωπαϊκά όργανα όταν υπάρξουν παράπονα από ένα φυσικό πρόσωπο ή από μία οργάνωση ε, ζήτησα από τον πρόεδρο της Επιτροπής να υποβάλει ένα νέο ερώτημα στην ε, νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου σχετικά με αυτό ώστε να λυθεί και η τελευταία αμφιβολία που μπορούσε να υπάρχει ε, μη υποστεθεί κάποιο νομικό θέμα. Και νομίζω ότι αυτό θα μας βοηθήσει σε σχέση με τις τροπολογίες, επαναλαμβάνω, που αφορούν στα τρία θέματα. Στο ρεζίστρ, στον ετήσιο έλεγχο και στην περίπτωση που υπάρξουν διαμαρτυρίες ή παράπονα ότι ένα κόμμα δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ή δεν είναι δημοκρατικό κόμμα με βάση τους κανόνες και τις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει βεβαίως στο τέλος, όπως είπαμε κύριε Πρόεδρε, να αποφασίσουμε πότε θα ψηφίσουμε. Πιθανόν να μπορούμε να το κάνουμε στις 11 του μηνός Θέλω να ακούσω και τις απόψεις ε, όλων των άλλων συναδέλφων. Ε, δεν θέλω να κάνω περισσότερα σχόλια. Έχουμε στείλει το, την πρόταση αυτή με τις τροπολογίες στους ε, Σάντου αλλά και σε όλους τους συναδέλφους. Και επομένως μπορούμε να συζητήσουμε επ' αυτών και για την κάθε μία χωριστά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Non mi pare, c'è qualcuno che vuole intervenire ancora una volta. Δεν νομίζω ότι θέλει κανεί να λάβει το λόγο ξανά για το θέμα των πολιτικών κομμάτων. Α, μάλιστα, κύριε Σντάφ. Παρακαλώ, κύριε Σντάφ. Σύντομα, επί της ε, διαδικασίας, νομίζω ότι πρέπει να ψηφίσουμε τη θέση μας το συντομότερο δυνατόν γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί τριμερής διάλογος και αρκετά εντατικός, από ό,τι φαντάζομαι, με το Συμβούλιο. πριν φτάσουμε σε μία ε, συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Νομίζω ότι η κυρία Γιαννάκου έχει παρουσιάσει πολλές συμβιβαστικές τροπολογίες για τις οποίες την ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλες πηγαίνουν προς τη σωστή κατεύθυνση. Υπάρχουν Ωστόσο, κάποια ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν περαιτέρω, κάτι το οποίο μπορεί να επιληθεί νομίζω μόνο με ψηφοφορία. Όπως για παράδειγμα το κατόφλι ένα τρίτο, ένα τέταρτο, ένα πέμπτο ε, των κρατών μελών ε, ως κριτήριο για την ίδρυση ευρωπαϊκών ε, πολιτικών κομμάτων. Γιατί υπάρχει διάσταση απόψεων επ' αυτού. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε να συμβιβαστούμε ως προς αυτό, νομίζω ότι πρέπει απλώς να ψηφίσουμε. Υπάρχει και το σημαντικό πρόβλημα της εφαρμογής. Ο μηχανισμός δηλαδή που θα διαλέξουμε για την εφαρμογή του νέου βελτιωμένου καθεστώτος πολιτικών κομμάτων. Γνωρίζουμε ως προς αυτό ότι υπάρχουν διαφωνίες ε, και εντός της Επιτροπής μας αλλά και μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε σχέση με το πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι η παράγραφος 2 του άρθρου 291 της συνθήκης ε, δίνει τη δυνατότητα στην Επιτροπή να εφαρμόσει τους κανονισμούς της Ένωσης και το να αποκόψουμε πλήρως την Επιτροπή από την οργάνωση της εφαρμογής του καθεστώτος είναι κατά την άποψή μου κάτι που θα ε, προκαλέσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά ενδεχομένως και, στο Συμβούλιο θα, θα οδηγηθούμε σε ε, ανεπίλητα νομικά προβλήματα. Θα ήθελα λοιπόν ε, να περάσουμε στην ψηφοφορία όσο το δυνατόν πιο σύντομα, για να μπούμε στον τριμερή διάλογο, ο οποίος θα διευκρινίσει ε, όλα τα ε, περιττέρω προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και κύριε Γιαννάκο. Εδώ έχουμε τρία διαφορετικά επίπεδα στα οποία θα ήθελα να σχολιάσω όσα μας είπε η κυρία Γιαννάκο. Πρώτα πρώτα. Λογικό είναι. Πριν ψηφίσουμε να διασκεδάσουμε τις αμφιβολίε που τυχόν έχουμε σε σχέση με το να προσφύγουμε δηλαδή στην νομική υπηρεσία για αυτά τα οποία μπορούμε να κάνουμε και για το, τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Οπότε και γι' αυτό ε, να μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα όρια αυτών των ε, αλλαγών που θέλουν να επιφέρουμε στα όσα ισχύουν. Στο καθεστώς δηλαδή για τα κόμματα πρώτα-πρώτα ακριβώς και σε σχέση με το Συμβούλιο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται, τι μπορούμε να αλλάξουμε και τι δεν μπορούμε και άρα για το τελικό αποτέλεσμα μόνο καλό μπορεί να κάνει το να διαπιστώσουμε αυτά τα όρια των δυνατοτήτων μας. Ε, δεύτερο θέμα, δεύτερο επίπεδο. Δεν ξέρω εάν αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι ο πυρήνας της μεταρρύθμισης που θέλουμε να γίνει. Πάντως ε, σίγουρα αυτό το οποίο αναφέρθηκε είναι η ουσία των διαφορών μας, των διαφορών που πρέπει να πω συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή. Θα πρέπει επομένως να προσπαθήσουμε να λιάνουμε αυτές τις διαφορές, να τις απαλείψουμε όπου έχουν σημασία. Εγώ πιστεύω ότι η διατύπωση αυτών των συμβαστικών τροπολογιών είναι μια διατύπωση που είναι πάρα πολύ θετική. Όχι δηλαδή το Γενοβούλιο απλώς διαπιστώνει ότι ε, όταν ένα κόμμα θέλει να καταστεί Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα ή Ίδρυμα το κατά πόσον επομένω πληρεί τις αντικειμενικές προποθέσει οι οποίες θεσπίζονται από αυτό το καθεστώς. αυτό είναι κάτι το οποίο το ονομάζουμε πιστοποίηση, διαπίστωση τέλο πάντων ότι πληρούνται κάποιε προποθέσει. Οπότε Έχουμε σχεδόν αυτή την ετησία αναθεώρηση των όσων διέπουν τη λειτουργία ιδρυμάτων και κομμάτων και τώρα κατά τρίτον και αυτό είναι το πιο επιμόχο θέμα ότι πάντοτε υπάρχει κάποια τελική απόφαση από πλευρά του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου όσον αφορά τη θεωρή περίπτωση κατά την οποία ένα Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα έρχεται σε ρήξη με τις βασικές αξίες. Αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι ε, ενσωματώνονται στη χάρτα των δικαιωμάτων. Ή τέλο πάντων το πούμε ευρύτερα, πιο αφηρημένε αξίε που ασπάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε θα πρέπει να διαπιστωθεί πρώτον ότι οποιοδήποτε Ευρωπαίος ή Ίδρυμα μπορεί να προβεί στη διαπίστωση ή καταγγελία τέτοιο μη σεβασμό αυτών των ε, αξιών. Επίσης ότι είναι δυνατόν η απόφαση να συζητηθεί από τα τρία θεσμικά όργανα, Συμβούλιο, Κομισιόν και Κοινοβούλιο και ότι επίσης είναι δυνατόν να συγκροτηθεί κάποιος φορέας, κάποιο όργανο που θα παρτίζει από κάποιους σοφούς οι οποίοι θα αποφαίνονται αφού ακούσουν τους εκπροσώπους αυτού του πολιτικού κόμματος που κατηγορείται. Και τελικά το θέμα θα αναπευθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το οποίο εκείνο θα είναι αρμόδιο να αποφασίσει, οπότε και έτσι θα έχουμε κάποιο είδου δικαστική προστασία μέσω κάποιων μηχανισμών που θα πλαισιώνεται από Κοινοβούλιο, Επιτροπή, κατόπιν επομένω γνωμοδότηση κάποιων αρμοδίων, κάποιων θα έχουν επιλεγεί γι' αυτό. Δεν ξέρω τώρα εάν ε, αυτό θα αποτελέσει την αποκρισταλωμένη θέση μας, αλλά νομίζω ότι έχουν τα πράγματα το σωστό δρόμο, τόσο να εμορφωθεί μια συνένεση μεταξύ εκείνων οι οποίοι στην Επιτροπή μας θα ήθελαν αυτή η απόφαση ε, τελικά αναλαμβάνεται από ένα δικαστικό όργανο. Τώρα, όσον αφορά το τρίτο θέμα, δηλαδή το, το πότε θα ψηφίσουμε, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Ντάφ. Το πιο σωστό είναι να αρχίσουν το νωρίτερο δυνατόν οι διαπραγματεύσει, ούτω ώστε να γνωρίζουμε ποια είναι η θέση του Συμβουλίου. Γιατί αλλιώ γυρίζουμε γύρω από τα ίδια και τα ίδια. Περιμένει το Συμβούλιο, περνάει ο καιρό και οι εκλογές του 2014 πλησιάζουν. Γι' αυτό νομίζω το πιο λογικό είναι να ψηφίσουμε νωρίες. Άλλωστε, το να ψηφίσουμε εμείς δεν σημαίνει ότι έτσι μορφώνονται οριστικά τα πράγματα. Έτσι κι θα γίνουν διαπραγματεύσεις. Οπότε καλύτερα να γνωρίζουμε τι πρεσβεύει η άλλη πλευρά. Όσο γίνεται νωρίτερα. Κύριε Ταρκόσκη. Α, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη. Συμπαθάτε με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 Μία από τις τροπολογίες αναφέρει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λειτουργεί βάσει αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, αναφέρεται στο άρθρο 10 της συνθήκης. Εγώ το κοίταξα αυτό το άρθρο και στην παράγραφο 3 λέει ότι κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να συμμετέχει στη δημοκρατική ζωή, στο δημοκρατικό βίο της Ένωσης. Δεν αναφέρεται τίποτε ε, σε σχέση με ε, τις αξίες ε, τι οποίε πρέπει να συμμερίζεται η πολιτική τάξη. Το κατά πόσο θα πρέπει να αναγνωρίζεται, να χρηματοδοτείται ένα πολιτικό κόμμα ε, από την Ένωση ε, είναι σχεδόν ε, δικαστικές αποφάσεις και όπως ε, αναφέρεται το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο θα έπρεπε να λάβει την τελική απόφαση. Όμως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι ένα δικαστικό σώμα, είναι ένα σώμα πολιτικό και η ιδέα ότι κάποιοι πολιτικοί θα αποφασίσουν κατά πόσο τα δικαιώματα ε, πρέπει να ε, την χάνουν σεβασμού ή στέρησης είναι κάτι το πραγματικά αδιανόητο. Κοιτάξτε, εγώ θα χαιρόμουν όλος ιδιαίτερος να αν υπήρχε ε, ισότητα των δύο φίλων και αν επιλειόταν όντως το ζήτημα αυτό στο πλαίσιο των πολιτικών κομμάτων ε, και μάλιστα χωρίς ιδιαίτερο προγραμματισμό. Αν όμως υπάρχει κάποιο είδους νομοθεσία θα πρέπει να υπάρχει και ένα κριτήριο επιλογής για ε, την ισότητα μεταξύ των φύλων λέτε ότι άλλα σημαντικά ζητήματα, πολύ πιο ε, σημαντικά ζητήματα στο πλαίσιο της επιλογής όπως για παράδειγμα η πολιτική πεποίθηση ε, ε, πρέπει να μην λαμβάνονται υπόψη ή άλλα να υπερισχύουν αυτόν. Για τη συμβιβαστική τροπολογία αντί τώρα λέτε ότι το κόμμα θεωρείται υπεύθυνο και ενδεχομένως να θα πρέπει να είναι υπόλογο των ε, μελών του. Για, για πόσα μέλη όμως μιλάμε. Μιλάμε για την πλειοψηφία των μελών ή μπορεί να είναι μόνο ένα μέλος. Το 2003 έγινε μια επιχείρηση απαγόρευσης ενός πολιτικού κόμματος ε, ε επί της βάσεως ε, κάποιων δηλώσεων ε, ορισμένων από το μελών τους και το ε, συνταγματικό δικαστήριο το οποίο ε, επρόκειτο να δεχθεί την αίτηση για τη δημιουργία του κόμματος αυτού, τελικά είπαν ότι όχι, δεν γινόταν κάτι τέτοιο, ότι δεν ήταν δυνατόν ε, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι να αποτελέσουν τμήμα πολιτικών κομμάτων. Για ποιο λόγο λοιπόν προτείνεται κάτι τέτοιο. Καταρχήν, να ευχαριστήσω τη Μαριέτα για τις συμβιβαστικές. Νομίζω το σημαντικότερο από όλα είναι να συμφωνήσουμε επί των αρχών. πρώτων, δηλαδή να είναι πιο ορατά τα ευρωπαϊκά κόμματα στην ε, πολιτική διαδικασία και να ρυθμίσουμε θέματα χρηματοδότησής τους και συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκές εκλογές, δημοψηφίσματα κλπ. Και τέλος όλη τη διαδικασία της καταχώρησης και επαλήθευσης γιατί αυτά είναι τα πιο επίμαχα θέματα. Νομίζω πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση και επιτρέπουμε η διαδικασία αυτή να αποπολιτικοποιηθεί, από κομματικοποιηθεί και να υπάρχει δυνατότητα να μην είναι μόνο ένα πολιτικό παιχνίδι, αλλά να αποφαίνονται και η δικαστική εξουσία συμφωνώ με τον Άντριο Ντάφ ε, ότι θα πρέπει να ψηφίσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα αφού διευκρινίσουμε κάποια θέματα με την νομική υπηρεσία αν και δεν ξέρω αν θα λυθούν τα προβλήματα που έχουμε. Γιατί πρέπει να υπάρξει ε, γνωμοδότηση της Επιτροπής το ταχύτερο δυνατόν. Όταν λοιπόν συμφωνήσουμε με τη φιλοσοφία της όλης προσέγγισης και τις σχετικές τροπολογίες, δεν νομίζω ότι έχει νόημα να κάνουμε κι άλλη και άλλη και παράλληλη συζήτηση και συμφωνώ με τον κύριο Νταφ ότι με την ψηφοφορία μόνο θα λυθούν ορισμένα επιμέρους πρακτικά θέματα για τη διαδικασία μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σόλτς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συμφωνήσω με όσους ζήτησαν γρήγορη διαδικασία σε ό,τι αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής μας σχετικά με τον κανονισμό. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Είναι τρεις βασικές θεματικές. Πρώτον, καταχώρηση. Δεύτερον, έλεγχος. Και ε, ένταξη, αποχώρηση ε, πολιτικών κομμάτων ευρωπαϊκών και σε ποιο βαθμό ε, ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που πρέπει να έχει ένα Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα. Και βεβαίως η συμμετοχή τους στις εκλογές. Επίσης, ε, δεν συμφωνώ με την ε, συμβιβαστική Α να περιορίζεται στις εκλογές ένα ευρωπαϊκό κόμμα, το οποίο είναι ένα συνασπισμός είτε εθνικών κομμάτων και ή μελών, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να συμμετέχουν στην διαδικασία περαιτέρω ολοκλήρωσης της Ένωσης. Άρα πρέπει καταρχήν να έχουν τη δυνατότητα σε ένα ευρωπαϊκό πολιτικό κόμμα να συμμετέχουν στα πολιτικά δρόμενα και όχι μόνο να ε, βλέπουμε ένα τέτοιο κόμμα σαν ε, προεκλογικό μηχανισμό. Πρέπει λοιπόν να μείνουμε στην αρχική αναφορά στο Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα, όπως αναφερόταν στο κείμενο της Κομισιόν. Τώρα, για την ε, καταχώρηση και τον έλεγχο ή την επαλήθευση των δραστηριοτήτων των Ευρωπαϊκών Πολιτικών Κομμάτων, ε, μετά την τελευταία συναντήση των σκιωδών, ε, έδωσα μια θέση δική μου και εξήγησε τις τροπολογίες μου και θέλω και εδώ στους συναδέλφους να πω στην Επιτροπή ότι πιστεύω ότι πρέπει να επιλέξουμε την απλούστερη οδό. Είναι μια διοικητική διαδικασία, είναι μια καταχώρηση και δεν είναι ε, διαδικασία πολιτικής αναγνώρισης των κομμάτων αυτών. Δηλαδή κάποια διεύθυνση, η Γενική Γραμματεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσε να επιφορτιστεί με κάτι τέτοιο και εκεί θα εξετάζονται τυπικά ε, τα έγγραφα που θα υποβληθούν. Αν, είναι, αν επιβεβαιωθεί η πληρότητα των εγγράφων αυτών, τότε το πολιτικό κόμμα θα καταχωρίζεται και νομίζω ότι αυτή είναι και η μοναδική τεχνική διαδικασία. Και έτσι ανταποκρινόμεθα και στα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι ο κάθε πολίτης, ε, κάθε πολίτης μπορεί να ε, προχωρήσει η συγκρότηση πολιτικών κομμάτων μαζί με άλλους και να συμμετέχει στη διαμόρφωση της ε, πολιτικής άποψης στην ε, πραγματικότητα κάθε χώρας. Κάθε Αυτό πρέπει να παραμείνει μια υπέρτατη αρχή που εμείς θα πρέπει να τηρούμε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και κατά την ε, επανεξέταση review των κομμάτων θα πρέπει να πω ότι και τα τρία θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είναι σε θέση να προβαίνουν στον, ε, στην αμφισβήτηση του ελέγχου αυτού, αλλά σε τελευταία ανάλυση η απόφαση για την ομιμότητα της δράσης ενός Ευρωπαϊκού Πολιτικού Κόμματος ε, θα πρέπει να μείνει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ε, ώστε να υπάρχει διαφάνεια και να είναι και κατανοητές ε, οι διαδικασίες μας ε, στους πολίτες, εις ό,τι αφορά το νομότυπο της δράσης των κομμάτων. Τέλος, δύο παρατηρήσεις που αφορούν, νομίζω, την τροπολογία G, τη συμβιβαστική G. για τα κόμματα που είναι μέλη και τα μεμονωμένα μέλη. Και αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί ένα κόμμα μέλος ή ένα συνδεδεμένο κόμμα ενός ευρωπαϊκού ή ένα... Μπορεί να, είναι, μπορεί να είναι πάρα πολλά τα κόμματα τα οποία είναι συγγενή προς ένα ευρωπαϊκό ε, πολιτικό κόμμα. και θα πρέπει να το διαφοροποιήσουμε σε σχέση με την ε, ε, ιδιότητα ενός μέλους, ενός ε, μόνο προσώπου. Ε, πρέπει να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Επίσης, για τη χρηματοδότηση και την επιστροφή χρημάτων ή την κάλυψη χρημάτων για προεκλογικέ εκστρατείες, νομίζω ότι ε, υπάρχουν ορισμένες, ε, ορισμένοι περιορισμοί και μη παραδεκτές διαδικασίες από το 86. Δηλαδή αυτό το θέμα της χρηματοδότησης νομίζω από το, από το 86 υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τη χρηματοδότηση. Ε, πρέπει λοιπόν όταν περιγράφουμε την επιστροφή δαπανών από προεκλογική εκστρατεία εδώ πρέπει να το αλλάξουμε και να επιτρέψουμε μια άλλη διατύπωση του κειμένου που θα ε, επιτρέπει την ε, ισοδύναμη συμμετοχή ευρωπαϊκών κομμάτων σε προεκλογικές εκστρατείες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίλαντ, ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι σύντομος. Θέλω κι εγώ γρήγορη διαδικασία, ταχεία διαδικασία. Βλέπω όμως ότι ε, είναι 400 περίπου οι συμβιβαστικές και οι συμβιβαστικές ε, καλύπτουν 89. Ε, υπάρχουν πολλές λοιπόν που παραμένουν, πολλές τροπολογίες που δεν καλύπτονται από τις συμβιβαστικές και θα πρέπει κάθε συνάδελφος ε, να έχει τη δυνατότητα να τα μελετήσει όλα αυτά και να ξέρει πολύ καλά ποια θα είναι η θέση του. Εγώ θα περιοριστώ σε λίγες, πάω στην συμβιβαστική M, ε, αυτό το, ε, αυτός ο φορέας με τα τρία επίπεδα με δυσκολεύει λίγο. Ε, είναι σαν να είναι μια επιτροπή σοφών που θα αποφαίνεται. Εγώ νομίζω ότι τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να λένε ότι ε, πιστεύουμε ότι ε, κάποιο κόμμα παρεκτρέπεται προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά και προσφεύγουμε στο δικαστήριο. Δεν χρειάζεται δημόσια κατακραυγή, ούτε χρειάζεται να ε, ασχοληθεί ιδιαίτερα. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένας φορέας λίγων με συμμετοχή ίσως και από τα ε, κόμματα τα οποία θίγονται. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να ζητήσουμε εδώ τμηματική ψηφοφορία για αυτήν. Στο σημείο Π, ε, η συγγήτρια που την ευχαριστώ πολύ, στο σημείο Π κάποιο πράγμα μου φαίνεται ότι δεν επαρκεί. Και σε, άλλους, ε, σε άλλες τροπολογίες είχα πει ότι αν έχω, αν επιστρέφονται αχρεωστήτως καταβληθέντα, βεβαίως ισχύει ο δημοσιονομικό μας κανονισμό. Αλλά η πραγματικότητα ποια είναι, ότι κάτω από ε, ορισμένες προϋποθέσεις και συσχετισμούς κόμματα που ζητούν κάτι παίρνουν χρήματα από κάποιους άλλους, διότι βεβαίως η πίτα είναι περιορισμένη. Και αν διαπιστωθεί ότι ένα κόμμα αδίκως ε, έλαβε ένα ποσό, τότε... Ε, δεν μπορεί να εξαφανιστούν τα χρήματα αυτά κάπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά νομίζω ότι είναι σωστό να ε, ξαναγυρίσει στο, στην πίτα που προβλέπεται για τα ευρωπαϊκά κόμματα, ούτω ώστε νομοτύπος, ε, τα, τα νομότυπα κόμματα να αξιοποιήσουν τα χρήματα τα οποία τους αφαιρέθηκαν, τα οποία είχαν στερηθεί. Ε, στην ΑΣ και την Ι νομίζω ότι εδώ ε, είναι λίγο ε, αδύνατο το κείμενο, η H ε, καλύπτει την τροπολογία μου για minimum democratic standards, ελάχιστα δημοκρατικά πρότυπα που να τηρούνται, αλλά αναφέρεται επίσης σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Λες και δεν γνωρίζουμε ότι σε αρκετά κράτη-μέλη σε πολλά επίπεδα υπάρχουν πολλές δυσκολίες. Όχι μόνο στο α ή β κόμμα, αλλά καμιά φορά σε όλα τα κόμματα. Όταν μιλάμε λοιπόν, ε, ε, όταν λέμε ελάχιστα πολιτικά ε, πρότυπα, φοβούμε ότι η μέχρι τούδε κατάσταση θα θεωρηθεί ως ελάχιστο αποδεκτό πρότυπο και δεν κάνει. Δεν πρέπει να μείνουμε στο σημείο που είμαστε. Πρέπει να ζητήσουμε περισσότερα πράγματα, καλύτερα πράγματα. Και στην συμβιβαστική τροπολογία Ή e, θα δούμε, γιατί αν είναι τόσο γενικόλογη, δεν, δεν μας δίνει κάτι συγκεκριμένο. Είτε λοιπόν θα κάνουμε το βήμα και θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι στη διατύπωση και βέβαια εδώ είμαι πολύ επιφυλακτικός, αλλά δεν μου αρέσουν οι γενικολογίες που δεν θα οδηγήσουν σε τίποτα ή θα οδηγήσουν σε κάτι πολύ υπερβολικό. Τέλος για το α, τη συμβιβαστική α, ε, μάλλον συμφωνώ με τον συνάδελφο Σόλτς πρέπει να πω. Τα κόμματα βεβαίως θα πρέπει να κατεβαίνουν σε προεκλογικές εκστρατείες να ε, προβάλλονται ε, τα κόμματα αυτά με τη συμμετοχή των πολιτών. Αλλά θα πρέπει να δούμε πότε αρχίζει το σημείο που θα πει το κόμμα ότι σε 10 κόμματα έχουμε φτάσει σε σημείο που μπορούμε να συμμετέχουμε και να έχουμε παρουσία στις ευρωπαϊκές εκλογές. Θα πρέπει πριν από κάποιους μήνες να έχουν ε, κάνει τη σχετική δήλωση. Δεν φτάνει. Ποιο θα είναι το χρονικό διάστημα. Θα, θα πρέπει δηλαδή ο πύχης να μην είναι πολύ υψηλό Και θα πρέπει να δούμε πότε είναι το σημείο που περνά κανείς το ρουβίκονα. Αυτό συμβαδίζει και με την ε, τροπολογία μου που λέει ότι είτε υπάρχουν εντολές είτε όχι, εάν ε, συμμετέχουν στις εκλογές θα πρέπει να ε, γίνεται μια διανομή των εδρών μεταξύ εκείνων που ε, κλαίγονται στο κοινοβούλιο. Ναι, e- Σα ευχαριστούμε. Κύριε Άγνιο, στήσε το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Σε σχέση με τη χρηματοδότηση και τη συγκρότηση των ε, ευρωπαϊκών κομμάτων, το δεν θα γίνει από τους φορολογουμένους. Και θυμάμαι τι έγινε τότε στην παλιά μας απικία. Τη είπα, λέγανε να μην υπάρχει φορολόγηση χωρίς εκπροσώπηση. Και εμείς ε, θέλουμε τώρα αυτό να κάνουμε, αυτό να πούμε στους φορολογούμενους. Θα σπάρουμε τα λεφτά να κάνουμε πολιτικά κόμματα, αλλά δεν δεχόμαστε κάποιες από τις απόψεις Μόνο θέλουμε τα λεφτά σας. Δεν θέλουμε τις απόψεις Αυτό δεν γίνεται. Ποιος θα ορίσει τι είναι ακραίο πολιτικό κόμμα κάποια ένωση πολιτικών προσώπων, πάντοτε κάποιος μέσα σε αυτήν έχει ε, κάποια ε, ακραία άποψη. Οπότε τι γίνεται, τότε θα, θα του βάζουμε την κόκκινη κάρτα, αυτό είναι μια κατηφόρα. Όχι, δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Θα πρέπει να μην σούμε χρήματα θα πρέπει τα ίδια τα κόμματα να αυτοχρηματοδοτούνται. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τελευταία πανέβαση και από τον κύριο Χέφνερ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε έγκαιρα στη λήψη αποφάσεων και σε οριστική επεξεργασία του καθεστώτος των κομμάτων. Πρέπει όμως το δίκαιο που θα θεσπίσουμε πρέπει να είναι καλό. Βλέπω ότι πολλές φορές έχουμε διαφορετική εικόνα του κόμματος, ενός κόμματος και της ε, ε, ελευθερίας των εκλογών, αν θέλετε. Τι σημαίνει η ελευθερία ε, των εκλογών και δημοκρατία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στην τάξη της κόρης μου εκλέγονται εκπρόσωποι της τάξης. Αγόρια, κορίτσια. Και φαντάζομαι ότι θα μπορούσε κανείς ε, να καταλήξει το παράδοξο να μπορεί να ε, βάζει υποψηφιότητα ένας εκπρόσωπος, ένας μαθητής για εκπρόσωπο, όποιος είχε επιτύχει σε προηγούμενες θητείες. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τα κόμματα δεν είναι μορφώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή άλλων θεσμικών οργάνων της Κομισιόν δημιουργούνται ελεύθερα. Δεν τα καθοδηγούμε εμείς για να σχηματιστούν τα πολιτικά κόμματα. Εμείς είμαστε οι υπεύθυνοι και κατευθύνουμε τα κόμματα που υπάρχουν, αλλά αν σχηματιστεί ένα καινούριο κόμμα, αυτό το κόμμα θα το φτιάξουν κάποιοι πολίτες που θα, θα συνασπιστούν και θα πούνε έχουμε κοινούς στόχους, κοινά ιδεώδη και θέλουμε να τα προωθήσουμε. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σημαντικό το καθεστώς του πολιτικού κόμματος να μην το περιορίσουμε με βάση τα κόμματα τα οποία δραστηριοποιούνται ήδη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή στα Εθνικά Κοινοβούλια. Δηλαδή να μην εξαρτήσουμε το καθεστώς από την επιτυχία ε, ήδη υφισταμένων, αλλά να πούμε ότι όπου συνασπίζονται πολίτες και πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, δηλαδή όταν είναι παρκής ο αριθμός των κρατών μελών, και υπάρχει ε, καταστατικό, δημοκρατικές ε, διαδικασίες, ε, οργανωτικές δημοκρατικό πρόγραμμα κλπ. Σε όλε αυτέ τι περιπτώσει θα πρέπει να επιτρέπονται και να θεωρούνται ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα. Το λέω αυτό με βάση τις τροπολογίες μου, 89 και 93, αλλά όχι μόνο, πολλές άλλες τροπολογίες συναδέλφων έχουν υποβληθεί και που ε, υποτίθεται ότι καλύπτονται από τη συμβιβαστική C, αλλά δεν βλέπω ουσιαστική τροποποίηση στην C, βλέπω μόνο μία διευκρίνηση στη συμβιβαστική C, ότι αυτό που ζητείτε εδώ για τα, τις οργανώσεις μέλη, μάλλον για τα συνδεδεμένα μέλη, ισχύει για τα ε, συνδεδεμένα affiliated parties, αλλά όχι για τη δεν, δεν αναφέρεται τίποτε άλλο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα που το σκαλίζουμε και το αναδεικνύουμε συνεχώς. Και όχι μόνο εμείς και η ομάδα μου και ο κύριος Σόλτς, ο συνάδελφος Βίλαντ και άλλοι πολλοί. Και θα ήμουν ευτυχής αν καταλήγαμε σε μια συμβιβαστική λύση εδώ. Συμβιβαστική όμως δεν σημαίνει την επανάληψη της αρχικής άποψη. Η συμβιβαστική είναι μια ε, τροπολογία που λαμβάνει υπόψη την άποψη των άλλων. Σε σχέση λοιπόν με το καθεστώς των κομμάτων θα πρέπει να καταλήξουμε συνενετικά, να πάψει να είναι τόσο επίμαχο θέμα αυτό ανάμεσά μας. Και λέω ειλικρινά ότι μέσα από τις συμβαστικές δεν φαίνεται προσέγγιση μεταξύ μας. Δηλαδή συζητούμε τι περιθώρια έχουμε για να κινηθούμε, αλλά δεν προσεγγίζουμε ένα τον άλλον. Σε άλλους τομεί όμως είναι αλλιώ τα πράγματα και υπάρχουν ε, θετικές ε, και ε, εξελίξεις που με χαροποιούν. Είναι σημαντικό να αποφύγουμε οτιδήποτε θα μπορούσε να ενισχύσει τις παρανοήσεις και να θεωρηθεί ότι τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα είναι κόμματα τα οποία καθοδηγούνται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Γι' αυτό είναι σημαντικό και αυτό που είπε ο κύριος Βίλαν, πολύ σημαντικό. Δεν νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να κρίνουμε τις ε, ε, οργανώσεις ε, τις ανταγωνιστικές με μας θα πρέπει ένα δικαστήριο να κρίνει ένα καταστατικό. γιατί αν η απόφαση επαφίεται σε μας έχω μεγάλο πρόβλημα και αμφιβάλλω αν οι ενδιαφερόμενοι και η κοινή γνώμη και οι ψηφοφόροι μας ε, θα μας αναγνωρίσουν την ουδετερότητα και την αμεροληψία που ζητείτε για κάτι τέτοιο. Διότι η δικαιοσύνη παρουσιάζεται παντού τυφλή και σε τέτοια επίμαχα θέματα ε, θα πρέπει να γίνεται ε, απονομή της δικαιοσύνης με τρόπο ουδέτερο αλλά και από έναν φορέα ουδέτερο. Εδώ θεωρώ ότι η τρίτη εξουσία ε, θα πρέπει να αναλάβει και όχι το κοινοβούλιο διάκριση των εξουσιών. Αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα που νομίζω ότι θα πρέπει να προσεγγίσουμε ο ένας τον άλλον και να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές λύσεις, ούτως ώστε πράγματι γρήγορα και συνενετικά να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε στο θέμα αυτό. η κυρία Γιαννάκου ε, για να απαντήσει. Ανησυχώ με το χρόνο μας, αν προλαβαίνουμε. Πρέπει να δούμε, ε, θα πρέπει να ψηφίσουμε άμεσα ε, και σε σχέση με το Συμβούλιο. 11 είπαμε την πρώτη ψηφοφορία. Πείτε μας εσείς τι γνώμη έχετε κυρία Γιαννάκου. Κύριε Πρόεδρε, θα αρχίσω από το τελευταίο σας σχόλιο ναι, μπορούμε να κάνουμε την ψηφοφορία στις 11 του μηνός στο Στρασβούργο, είναι Δευτέρα ή μπορούμε να την κάνουμε στις 14 που είναι Πέμπτη. Ένα, μια από τις δύο εναλλακτικέ λύσεις. Και νομίζω ότι πρέπει να την κάνουμε. Ε, τώρα, ως προς τα λεπτά σημεία της έκθεσης, κύριε Πρόεδρε, γιατί πραγματικά από τις τροπολογίες που γίνανε είναι φανερό ότι όλοι οι συνάδελφοι θέλουν να συμβάλλουν σε αυτή την έκθεση ότι έχει ενδιαφέρον δηλαδή για όλους και για τις πολιτικές ομάδες. Ε, παραδείγματος χάρη το να μνημονεύεται το να μνημονεύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα με λεπτομέρειες κλπ δεν χρειάζεται στο συγκεκριμένο άρθρο όπως αναφέρθηκε γιατί όταν αναφέρονται τα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στη συνθήκη είναι σαν να υπάρχουν όλα. Δεν υπάρχει καμία διαφορά. Δεύτερον, σε σχέση με τα, αυτά που είπε ο κύριος Βίλαν, οι τροπολογίες είναι σαφείς. Προβλέπουν το δικαίωμα και το έχει αυτό το δικαίωμα και το Κοινοβούλιο και η Κομισιόν και, και το Συμβούλιο να στείλουν κάτι στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, θέλω να το επαναλάβω πάλι, είναι όποιος διαμαρτύρεται για ένα κόμμα εμείς να το στέλνουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο διότι κινδυνεύουμε να στείλουμε ψεύτικες και γελίες καταγγελίες στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα screening, μία, μία άποψη. Τώρα ο κύριος Ντάφ παραδείγματος χάρη εδώ λέει εννέα μέλη να είναι τα eminent persons. Όμως ε, Άντριου όταν λέμε επιτροπή σοφών πάντοτε εννοούμε λίγους. Δεν εννοούμε τόσους πολλούς, εννοούμε πάντοτε λίγους κάποιους ανθρώπους σοβαρούς οι οποίοι θα, δώσουν μια, θα κάνουν μια σοβαρή γνωμοδότηση. Τα τρία σημεία που σας ανέφερα, όπως σας είπα έχουμε στείλει ερώτημα, ο πρόεδρος στέλνει ερώτημα στο, στη νομική υπηρεσία για το registration, το οποίο είναι τυπική υπόθεση, διοικητική, δεν είναι πολιτική υπόθεση για, το ετήσιο, για τον ετήσιο έλεγχο και κυρίως για αυτό το θέμα που μας έχει όλους απασχολήσει. Τι γίνεται αν κάποιος διαμαρτυρηθεί ότι ένα κόμμα δεν είναι δημοκρατικό, η συμπεριφορά των μελών του δεν είναι σωστή κτλ. Αυτό θα πάει στο δικαστήριο στο τέλος, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Επομένως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχούμε ότι δήθεν εμείς θα είμαστε μεροληπτικοί και να δημιουργηθεί θέμα. Τέλος, ως προς το τι είναι τα κόμματα. Βεβαίως τα κόμματα δεν τα καθορίζουμε εμείς, ούτε λέμε εμείς τι θα κάνουν. Λέμε όμως ότι για να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον εκλέξει ένα βουλευτή και να προέρχονται από το 1 τέταρτο των χωρών. Και εγώ εδώ επιμένω κύριε συνάδελφοι στο 1 τέταρτο των χωρών. Υπάρχουν προτάσεις το 1 τρίτο, το 1 πέμπτο κτλ. Βεβαίω μπορεί να κάνει όποιο θέλει κόμμα και α, είναι μέσα, μέσα στο δικαίωμά του ως Ευρωπαίος πολίτης. Αλλά όταν το κόμμα αυτό γίνεται θεσμός ο οποίος χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης τότε πρέπει να υπάρχουν κριτήρια. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν κριτήρια. Θα υπάρχουν προϋποθέσεις και κριτήρια. Και χωρίς αμφιβολία δεν είναι σωστό να χρηματοδοτηθούν κόμματα που δεν έχουν εκλέξει ποτέ κανέναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό δεν είναι λογικό. Επομένως ένα κόμμα μπορεί να κάνει registration στο Κοινοβούλιο αν δημιουργηθεί για πρώτη φορά και όταν θα εκλέξει τουλάχιστον έναν ευρωβουλευτή μπορεί να χρηματοδοτηθεί. Και αυτό ίσχυε και μέχρι σήμερα. Θέλω να πω κύριε Πρόεδρε ότι πολλά από αυτά ίσχυαν και μέχρι σήμερα. Δεν είναι πρωτοφανή η καινούρια. Νομίζω λοιπόν και εγώ ότι μπορούμε να ψηφίσουμε τις τροπολογίες συμβαστικές και ε, όλες τις άλλες στο Στρασβούργο. Εν τω μεταξύ, εγώ θα καλέσω τους ε, σκιώδεις να συναντηθούμε πάλι πριν από όλα αυτά. Έτσι, θα καλέσω πάλι τους σκιώδους εισηγητές μέσα σε αυτή τη βδομάδα εάν συμφωνείτε. Να τα πούμε άλλη μια φορά, να συνεννοηθούμε και νομίζω ότι μπορούμε να ψηφίσουμε στις 14 του μηνός του Στρασβούργου. Στις 11 του μηνός κύριε Πρόεδρε. Αν όχι στις 14 για να τελειώσουμε. Για να μπορέσουμε να αρχίσουμε τον τρίλογο όπως πολύ σωστά είπε ο Άντριο ε, να αρχίσουμε τη συνεννόηση με το Συμβούλιο όπου στο Συμβούλιο ξέρουμε που είναι τα λεπτά σημεία είναι αυτό με τα δημοψηφίσματα κλπ για ορισμένες χώρες ε, αλλά κύριε Πρόεδρε τώρα η, Ευρώπη είναι ένας χώρος ελεύθερης διακίνησης αγαθών υπηρεσιών προσώπων και κεφαλαίων. Ποιος εμπόδισε μέχρι σήμερα οποιονδήποτε Ευρωπαίο πολιτικό να πάει και να συμμετάσχει σε εθνικές εκλογές κτλ. Το θέμα είναι η χρηματοδότηση. Εκεί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Δεν ζητάμε περισσότερα χρήματα. Θέλουμε να αυξήσουμε τη διαφάνεια τη λειτουργικότητα και την αποτελεσματικότητα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Άρα, Δεν έχω ζητήσει άλλο το λόγο. Όσο από πλευρά διαδικαστική, η πρόταση τη κυρία Γιαννάκου είναι να κανονίσουμε πότε θα γίνει, αν συμφωνείτε, την ψηφορία να γίνει στι 11 Μαρτίου. Έτσι δεν είναι καλός. Εντάξει. Να δούμε μήπως κάτι άλλο προκύψει έκτοτε. πάντων, καταρχήν λέμε επομένω ότι ψηφορήθηκαν στις 11 Τρίτου. Εντάξει, συμφωνείτε, οπότε επομένω αυτό ε, οριστικά θα γίνει έτσι. Και τώρα προχωρούμε στο επόμενο θέμα που είναι το σημείο υπαριθμών 5, το οποίο αφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν ώψη των εκλογών του 2014 και έχουμε την ε, έκθεση των Γκουαλτιέρη και Ταρκόφσκι. Για να δούμε τώρα, να ακούσουμε τους ηγητές. Πρόκειται για την τελευταία συζήτηση του θέματος. Γιατί αύριο θα γίνει η ψηφοφορία. Ποιος από τους δύο συνεισηγητές θα ήθελε πρώτος να μιλήσει. Κύριε Τασκόσκη. Well, uh, what we... Αυτό που προσπαθήσαμε να υποβάλουμε είναι κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες ε, μέσω των οποίων κάποιες από τις ανησυχίες και κάποια από τα προβλήματα των συναδέλφων λαμβάνονται υπόψη. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε την ρεαλιστική μας πρόταση, οπότε αυτό δεν θα έπρεπε να εκπλήσει κανέναν. Το γεγονός δηλαδή ότι όλες οι τροπολογίες ε, σκοπό έχουν να αλλάξουν τη φύση της ε, πρότασής μας ε, απορρίπτονται εξ αρχής. Όσον αφορά επίσης τα επιχείρηματα που μεταβάλλουν κάποιες από τις λεπτομέρειες της πρότασής μας ε, όσον αφορά την κατανομή των εδρών ε, μεταξύ ε, των κρατών μελών εφόσον υπερασπιζόμαστε τη συγκεκριμένη πρόταση, θα βάλουμε μείον στον κατάλογο ψηφοφορίας στις συγκεκριμένες τροπολογίες. Και δεν έχουμε βεβαίως συμπεριλάβει συμβιβαστικές τροπολογίες αυτές τις απόψεις. Όσον αφορά όμως κάποιους γενικούς κανόνες, ε, καταλήξαμε ότι κάποιες από τις τροπολογίες πήγαιναν προς τη σωστή κατεύθυνση και επί της βάσεως αυτής έχουμε υποβάλει κάποιες συμβιβαστικές τροπολογίες. Απλώς να πω κάτι ε, σε σχέση με τη φόρμουλα. Ανεξαρτήτως του πιστεύουμε εμείς ε, για τις διάφορες μεθόδους, τις διάφορες φόρμουλες, ε, στην Επιτροπή μας ε, υπήρχε μία συμφωνία και άλλωστε αυτό είχαν ε, δείξει οι κάποιες που είχαν γίνει προηγουμένως, να μην έχουμε συγκεκριμένες φόρμουλες στο, στην, στην έκθεση της χρησιμοποιούμε στο σχέδιο εκθέσεως για να έχουμε μία βάση, αλλά δεν θέλουμε να αναφερθούμε συγκεκριμένα σε μαθηματική και ε, μεθόδους ε, στην τελική μας έκθεση και στις συμβιβαστικές τροπολογίες. Όσον αφορά τώρα τη σχέση με, την, ε, με ολόκληρη τη μεταρρύθμιση του θεσμικού συστήματος και τις έδρες, η άποψή μας είναι ότι αυτά τα δύο πράγματα πρέπει να συνδέονται και να αναφέρονται. Αν θέλουμε να έχουμε μια επαναστατική μεταρρύθμιση που να πηγαίνει πέρα από την ρεαλιστική μας προσέγγιση, θα πρέπει να έχουμε, θα πρέπει να σκεφτούμε μια πολύ ευρύτερη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών οργάνων στο μέλλον. Όσον αφορά τώρα ένα βιώσιμο σύστημα κατανομής εδρών για το μέλλον. Δεν σημαίνει ότι αυτό δεν θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη από κοινού με τη στάθμιση των δικαιωμάτων ε, ψηφοφορία στο Συμβούλιο. Είναι κάτι το οποίο αναφέρεται πολύ συχνά ε, στι τροπολογίε συναδέλφων. Ε, επίσης, η άποψή μας είναι ότι πριν από το τέλος του 2015 μια νέα πρόταση για το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο με σκοπό την εγκαθίδρυση συστήματος ε, ε, εγκαίρως για την, τον επόμενο ε, εκλογικό κύκλο. Πρέπει να, ληφθεί, πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο, πρέπει να υπάρχει ένα βιώσιμο ε, σύστημα και αυτό ήταν άλλωστε και επιθυμία πολλών συναδέλφων μας, ότι θα έπρεπε να στραφούμε προς το μέλλον και να το συζητήσουμε. Όσον αφορά τώρα τις ε, λεπτομέρειες, αποφασίσαμε επίσης να μιλήσουμε για τις αρχές της φθήνουσας αναλογικότητας χρησιμοποιώντας βέβαια ως σημείο αναφοράς ε, κάποιο από τον προβληματισμό που ήταν ε, πίσω από την έκθεση ε, Σεβερίν Λαμασούρ. Είναι άλλωστε και η δική μας συλλογιστική αυτή και χρησιμοποιώντας παραδείγματα και αποσαφηνήσεις των συναδέλφων μας. Και θα δείτε ότι αποφασίσαμε να μιλήσουμε λεπτομερώς για τις αρχές αυτές δανειζόμενοι κάποιε, κάποιων συναδέλφων, Χέφνερ, Διόν, Μπενέρ, ε, Τάραντ ε, ε, και κάποιες του Άντριου. Προσπαθήσαμε να πάρουμε πολύ σοβαρά όλες τις τροπολογίες οι οποίες δεν ε, αποδυναμώνουν ε, την ε, βασική κατεύθυνση της εκθεσής μας. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε συμβιβαστικές τροπολογίες που προετοιμάσαμε. Και εγώ και ο Ρομπέρτο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκολτιέρη. Σας ευχαριστώ. έχω και πάρα πολύ να σας προσθέσω. Γενικώ, πάντως, πρόκειται να παρουσιάσουμε μια σειρά τροπολογιών. Γιατί όπως είπαμε την τελευταία ώρα που τα συζητήσαμε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ ε, σημαντικές προτάσεις. Οπότε και αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε είναι να καλύψουμε όσο γίνεται περισσότερε από αυτές και έτσι να δούμε πώς θα βελτιώσουμε το ψήφισμα. Ήδη ο συνάδελφος σας ε, είπε ποια είναι τα βασικά στοιχεία από τις βασικές προτάσεις, οπότε έτσι να μπορέσουμε να γίνει το μήνυμα πιο δυνατό όσον αφορά το ότι χρειάζεται μία πρόταση να διαμορφωθεί πρώτου τέλους του 2015. Όπως είπε ο Βίλαν και άλλοι όσον αφορά τον έχουμε κάποιο είδου βιώσιμο και διάφανο μηχανισμό. Την άλλη μεριά πάντως εδώ πέρα έχουμε και μια ευρύτερη πρόταση, μέρο τη οποία αποτελεί και η παρούσα το πώ θα γίνει επομένω ε, η ψηφοφορία, τι θα γίνει και στο Συμβούλιο, τι θα προβλέπει και η ψηφοφορία όσον αφορά κάποια αναθεώρηση τη συνθήκη που θα υποβληθεί από το Κοινοβουλίο στα πλαίσια τη ε, εντολή για μια ε, συντακτική συνέλευση που θα λάβει μέρο στο μέλλον. έχουμε την τροπολογία 38 του Χέφνερ και άλλου συναδέλφου. Ε, θα καλύψουμε το πρόβλημα του ε, ορισμού. Θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. θα μπορούσαμε να έχουμε έναν βιώσιμο κανονισμό και αυτό να ισχύει και για τον ίδιο αριθμό εδρών. ανεξάρτητα από την πρόταση που υπάρχει ε, του να αυξηθούν οι έδρε. Επομένω, ε, κατά κάποιο τρόπο, εδώ αναμειγνύουμε τη δική μα πρόταση και την πρόταση του κ. Χεύνερ και του άλλου συναδέλφου για να βελτιώσουμε το ψήφισμα. Αυτά όσον αφορά τι συμβαστικέ προτάσει. Και να δούμε κατά πόσο μπορούμε εδώ να δούμε κάποια πρόταση επί τη βάση ότι χρειάζεται να γίνει κάποια αναθεώρηση. Με δεδομένη την διαδικασία που ισχύει ότι ε, να δούμε πώς θα υπάρχει η ευρύτερη δυνατή πλειοψηφία που να συγκεντρώσει το κείμενο ή να δούμε κατά πόσο μπορεί να υπάρχει ομοφωνία για να στηρίξει στο Συμβούλιο. Και εμείς έτσι διατυπώσαμε την ε, πρότασή μας από τη βάση αυτών των αρχών, των τριών αρχών. Και είπαμε ότι έχουμε αυτή την ευθύνη αναλογικότητα σύμφωνα με την πρόταση αυτή. Οπότε και εμείς θα πρέπει να έχουμε το ελάχιστο και το μέγιστο κατόφλι και κατά συνέπεια διασκευάσει των προκνοφέτων των τριών αρχών να προβούμε σε την πρότασή μα των δύο φάσεων. Τι ξέρετε, πρώτα πρώτα δηλαδή, να εφαρμοστούν πλήρω αυτέ οι τρει αρχέ και στη δεύτερη φάση, στο δεύτερο στάδιο, να υπάρχει κάποιο πολιτική αντιστάθμιση, ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε μια λύση ρεαλιστική. Μια λύση που ακόμη θεωρούμε ότι είναι η λιγότερο κακή, η λιγότερο ατελής όχι ότι είναι η τελειωτέρα, αλλά λιγότερο ατελής και γι' αυτό το λόγο. Όταν ε, ερχόμαστε στο θέμα των στοιχείων, των αριθμών, είπαμε οι σχετικές τροπολογίες να απορριφθούν. Βεβαίω, να δούμε τι θα γίνει στην ψηφοφορία. Μπορεί κάποιες από αυτές τις τροπολογίες να περάσουν. Όμως, η δική μας πρόταση είναι να μείνουμε, να διατηρηθεί, να παραμείνει το αρχικό κείμενο. Ευχαριστώ. Θέλω να ρωτήσω του συνεισηγητέ αν ε, υπάρχουν οι τροπολογίες ε, υπομορφή σχεδίου για να τι δούμε και να έχουμε πιο καλή ανταλλαγή απόψεων. Δηλαδή κατάλαβα ότι δεν δέχεστε τροπολογίες που να αλλάζουν τον αριθμό των εδρών που κατανέμονται σε ε, κάποια χώρα, σε όλες τι χώρε. Αλήθεια είναι. Ακούστε, εμείς δεν έχουμε την αρμοδιότητα, την εξουσία να δεχτούμε ή να μην δεχτούμε τις τροπολογίες. Θα κάνουμε κατάλογο ψηφοφοριών του εισηγητή, οι πολιτικές ομάδες θα κάνουν τις δικές τους και μετά θα δούμε, μετά την ψηφοφορία δηλαδή, ποιες τροπολογίες θα γίνουν δεκτές και ποιες όχι. Εμείς προτείνουμε να μείνουμε στα ε, νούμερα που έχει η δική μας η πρόταση. Ωραία γιατί αν αποφανθούν από κοινού με τον ίδιο τρόπο το ΕΛΚ και οι σοσιαλιστές δημοκράτες, ε, τότε η πυθός τους αυξάνεται. Αυτό που θέλω συγκεκριμένα να ρωτήσω είναι το εξής. Υπήρξε τροπολογία του Άντριου Νταφ και άλλων. Συγκεκριμένα για το θέμα του να αφαιρεθεί από την Αυστρία μια έδρα και να μην μειωθούν οι έδρες της Σουηδίας. Θέλω να ξέρω τι πιστεύετε για την τροπολογία αυτή, πρώτον διότι βελτιώνει την φθήνουσα αναλογικότητα, ένα αυτό, και δεύτερον συνάδει και με την αρχή σας να παίρνετε μόνο μια έδρα από κάθε χώρα. Οπότε ξεπλάγει λίγο που δεν δεχτήκατε αυτή την τροπολογία και θέλω να ξέρω γιατί. Ακούστε. Θα πρέπει να τηρηθεί αυτός ο κατάλογος που έχουμε και γιατί υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σειρά με τις οποίες με την οποία έχει λόγο. Οπότε τώρα ο κύριος Νταφ, ο κύριος Φόξ. Είμαι ευγνώμων στις, ε, για τις εξηγήσεις των εισηγητών και είμαι βέβαιος ότι οι συμβιβαστικές τροπολογίες για τα επόμενα, ως, επόμενα, ως επόμενο βήμα θα γίνουν δεκτές από την Επιτροπή και σίγουρα από την, Επιτροπή των, από την ομάδα των φιλελευθέρων που θέλει να, πολύ να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό και να διαμορφώσουμε τη θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τις ε, μεταρρυθμίσεις που θέλει για το όργανο αυτό. Και θέλουμε και στο Συμβούλιο να προχωρήσει το θέμα και να δημιουργηθεί στο Συμβούλιο ε, ισχυρότερη ισορροπία στις ψηφοφορίες Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Και αν μπορούμε να αποφανθούμε σαφώς υπέρ της ανάγκης για ε, συνέλευση για τη μεταρρύθμιση της συνθήκης, ώστε να έχουμε ε, βιώσιμη λύση για όλα αυτά, τότε οπωσδήποτε θα χρειαστεί σύμφωνη γνώμη των φιλελευθέρων και εγώ περιμένω ότι θα υπάρξει ευρύτατη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο. Τώρα, για τους αριθμούς, τα αριθμητικά στοιχεία. Πάντοτε είναι δύσκολο να, πιο δύσκολο να φτάσετε γνήση υπέρ μιας βιώσιμης ρεαλιστικής λύσης από τη μια, θέση επί των αρχών. Πάντως ε, είδα ο μπίνακα για το σημείο 3 Νομίζω κάποια στοιχεία δεν μπορούν να γίνουν δεκτά. Η τροπολογία μας 44, για παράδειγμα, παραβιάζει τη συνθήκη. Και νομίζω ότι αυτό θα πρέπει ο πρόεδρος να το, αυτή την τροπολογία είναι τη απαράδεκτη. Επίσης, ε, για τους Ιρλανδούς συναδέλφους, που κάνουν ένα σωρό ευφυείς προτάσεις ε, για να ενισχύσουν την ε, Ιρλανδική αντιπροσωπεία. Με κάθε σέβας πρέπει να τους πω ότι και εκείνοι πρέπει να δεχτούν ότι η Κροατία και η Ιρλανδία θέλουν να έχουν τον ίδιο αριθμό βουλευτών Νομίζω ότι είναι δίκαιο και σωστό αυτό και αν το παραβιάσουμε θα έχουμε πρόβλημα όλοι μας. Τώρα, για το θέμα του κυρίου Φόξ και την ανομαλία ότι υπάρχει διαφορά δύο εδρών μεταξύ Ουγγαρίας και Σουηδίας. Για με διαφορά πληθυσμιακή μόνο 475.000. Νομίζω ότι αυτό όντως είναι λάθος και πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να υποστηρίξουμε τις σχετικές τροπολογίες και που είναι και αρκετές Κάποιες μάλιστα ποινικοποιούν τους Αυστριακούς παίρνοντάς τους μια έδρα, αλλά κάποιες άλλες τροπολογίες προσεγγίζουν το θέμα με τρόπο διαφορετικό. Και βλέπω ότι η τροπολογία 55 έχει αποσυρθεί που την είχαν υποβάλει Σουηδοί συνάδελφοι. Θέλω όμως να την βάλω πάλι, να την επανακαταθέσω εξ του κυρίου Φερχόφστατ. Ευχαριστώ πολύ. Α, ευχαριστώ, ο κύριος ε, Χέφνερ. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Πρόεδρε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Πρέπει να συνεννοηθούμε για δύο πράγματα εδώ. Πρώτον, ότι αυτή θα είναι η τελευταία περίπτωση κατά την οποία με σπροξήματα πάνω, κάτω, δεξιά και αριστερά πάμε να βρούμε μια λιγότερο ή περισσότερο ικανοποιητική λύση, ενώ γνωρίζουμε ότι δεν ακολουθούμε διαφανείς και δίκαιους κανόνες, αλλά προσπαθούμε στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ε, εκφράσουμε την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας και μετά να κάνουμε διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και να δούμε τι θα βγει από αυτή τη διαπραγματευτική διαδικασία και το παζάρι ε, που ακολουθεί. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να συμφωνήσουμε καταρχήν ότι στο μέλλον χρειαζόμαστε έναν κανόνα ε, με βάση τον οποίο η κατανομή των εδρών θα εξαρτάται από το μέγεθος και τον πληθυσμό των κρατών μελών. Δηλαδή το πληθυσμό και το μέγεθος και θα είναι καθαρός κανόνας ξεκάθαρος ως αποτέλεσμα μιας μαθηματικής φόρμουλας που θα ακολουθεί την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας. Είναι δυνατό να γίνει αυτό και με βάση τις προδιαγραφές και επιταγές της συνθήκης. Έχουμε υποβάλει σχετική τροπολογία και πρέπει να πω ότι για μας η προθυμία, η ετοιμότητα να εξεταστεί μια πραγματιστική λύση, όχι η λιγότερο ικανοποιητική, εξαρτάται από το αν θα μπορέσουμε να συμφωνήσουμε ότι μετά την, τις επόμενες ευρωεκλογές θα συγκροτηθεί μια συνέλευση που και για άλλους λόγους χρειάζεται και η οποία θα εξετάσει τα θέματα αυτά και θα φροντίσει τους ώστε να υπάρχει βιώσιμη λύση διαφανής και δίκαιη για όλους. Και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε χρειάζεται μια ρεαλιστική λύση και η ομάδα μου και εγώ προσωπικώς συγκαταλέγομαι μεταξύ εκείνων που δέχονται την αρχή που πρόβαλαν οι Ρομπέρτο και Ράφαλ για αυτήν την ε, υπόθεση. Δηλαδή, εντάξει, αν πρόκειται για πραγματιστική προσέγγιση ε, που θα μας φέρει προσεγγιστικά πιο κοντά στο στόχο μας, τότε δεν θέλουμε να αλλάξουμε περισσότερη από μία έδρα προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε σχέση με τη σημερινή κατανομή. Εμείς ε, υποβάλαμε μια λίγο διαφορετική πρόταση γιατί στην ε, τροπολογία μας αυτή λέμε ότι ε, ως βάση θα χρησιμοποιήσουμε μια, ένα σαφή μαθηματικό τύπο που θα δώσει καθαρή κατανομή εδρών ε, των 751 ε, ε, εδρών μεταξύ των κρατών μελών με διαφορετικά ποσοστά και πάντοτε παρόλο που μπορεί να υπάρχουν διακυμάνσεις θα έχουμε καθαρά αποτελέσματα. Εμείς εφαρμόσαμε αυτό το μαθηματικό τύπο και λάβαμε υπόψη μας και την αρχή ότι κανένας δεν πρέπει να χάσει περισσότερο ή να κερδίσει περισσότερο από μία έδρα αυτά είναι θέματα ρεαλισμού για μας. Τι δηλαδή είναι το δυνατό και το εφικτό. Ο μακροπρόθεσμος στόχος για μας είναι ε, αυτός που ανέφερα στην αρχή και που είναι το πιο σημαντικό. Τώρα, για την τροπολογία μας 38 δύο λόγια, γιατί έχω την εντύπωση ότι δεν έγινε πολύ καλά κατανοητή. Αυτή η τροπολογία προέκυψε μετά από συζητήσεις με μαθηματικούς με τους οποίους ε, είχαμε μια αλληλογραφία. Και μάλιστα τα ακούσαμε αυτά και τα είπαν ξεκάθαρα και στην ακρόαση που έγινε εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός, τόσο μεγαλύτερο το δικαίωμά του για περισσότερες έδρες και όσο μεγαλύτερος ο πληθυσμός ενός κράτους μέλους, τόσο μεγαλύτερος ο αριθμός των κατοίκων που εκπροσωπείται από κάθε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, αυτό, αυτός ο συνδυασμός δεν μπορεί να υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Εμείς επιλέξαμε λοιπόν μια διατύπωση η οποία επιλέξαμε μια διατύπωση που δεν θα αντέξει στην περαιτέρω διαδικασία και μας το είπαν ότι δεν θα αντέξει. Παρακαλώ λοιπόν κατεπηγόντως και συμβουλεύω παρενώ να μην επιλέξουμε έναν ορισμό που δεν θα μπορέσουμε να τον τηρήσουμε στο μέλλον, να είναι ορισμός με διατυπωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να ισχύει και στο μέλλον. Γι' αυτό υποβάλαμε την τροπολογία 38 που λέει πριν στρογγυλέψουμε σε άρτιους αριθμούς, πριν από το στρογγύλεμα γίνεται. Α, α, το, α εντάξει, άμα έγινε δεκτό μη συνεχίσω. Υπάρχουν και άλλα, ε, κάποια τεχνικά θέματα, αλλά αυτό μου ήταν πολύ σημαντικό γιατί και σε ε, τυπικό επίπεδο και σε μαθηματικό επίπεδο μην μπούμε σε βάλτο, αλλά να μπορούμε να έχουμε κάτι που θα το υποστηρίξουμε και θα ισχύει και στο μέλλον. Ε, τώρα περιμένω τις συμβιβαστικές τροπολογίες βέβαια ως βάση για τις περαιτέρω συζητήσεις και προσβλέπω σε καλό αποτέλεσμα στο τέλος. Θα ήθελα απλώ να τονίσω ορισμένες ε, αρχές. Νομίζω ότι η ρεαλιστική λύση που βρέθηκε είναι λογική. Ακόμη και αν κάποιοι εξημών ε, που προερχόμαστε από κράτη-μέλη που ε, θα χάσουν μια έδρα, θα προτιμούσαν να μην χάσουν την έδρα αυτή, νομίζω όμως ότι στο πλαίσιο ενός πραγματικού ευρωπαϊκού πνεύματος πρέπει να ε, αναγνωρίσουμε ότι οι εισηγητές έχουν καταλήξει σε μια πολύ αποδεκτή λύση. Νομίζω ότι πρέπει και να εκπαιδεύσουμε κατά κάποιο τρόπο ε, την κοινή γνώμη μας ε, ότι αυτή είναι η καλύτερη λύση. Είναι μάλιστα καλύτερη και από τη λύση της ε, αύξησης των μελών, των εδρών, που επίσης θα ήταν μια ρεαλιστική λύση. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω, να υπογραμμίσω την προσπάθεια αυτή των συναδέλφων μας ε, Τσασκόφσκι και Γκουαλτιέρη. Θα ήθελα επίσης να πω ότι εγώ δεν πιστεύω στους μαθηματικούς τύπους, θα απογοητεύσω τους συναδέλφους ε, που τους αρέσει πολύ ο μαθηματικός τύπος, γιατί είναι το ευκολότερο πράγμα να προσαρμόσει κανείς ε, ή να, να εξεύρει ένα μαθηματικό τύπο για μια συγκεκριμένη κατάσταση. Αν ζητήσετε από ένα μαθηματικό να βρει ένα μαθηματικό τύπο για την ε, συγκεκριμένη λύση, για παράδειγμα, βεβαίως θα μπορέσει να το κάνει. Μπορούμε λοιπόν να τα υποστηρίξουμε όλα με ένα μαθηματικό τύπο και να τελειώνει η υπόθεση. Δεν είναι όμως αντικειμενικός ο μαθηματικός τύπος, γιατί εδώ συζητούμε πολιτικά και συνταγματικά προβλήματα. Δεν συζητούμε μαθηματικούς τύπους. Μπορούμε βέβαια να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε πιο διαφανή και πιο αντικειμενικά κριτήρια ίσως. Όμως τα προβλήματα θα παραμείνουν πολιτικά και συνταγματικά. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε αυτή τη διαφάνεια και την αντικειμενικότητα. Όμως ε, είναι γεγονός ότι είναι ένα μεγάλο πολιτικό πρόβλημα. Επίσης, κάτι άλλο. Δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με τους πληθυσμούς, αλλά και με τα κράτη. Και αυτό είναι ο λόγος, ε, γι, αυτό, για, γι' αυτό ακριβώς ε, έπρεπε να απαντήσω όπως απάντησα στην προηγούμενη παρέμβαση του κύριου Χέφνερ ο κανόνας της κατανομής. Ναι, εντάξει, αλλά εμείς δεν έχουμε ε, άλλο σώμα. Ένα μόνο σώμα υπάρχει, γιατί όταν υπάρχει δύο, όταν υπάρχουν δύο πρέπει κάπως να εξισορροπηθούν οι, ε, τα, οι αρχές. Και σας λέω, Αν μου πείτε ότι μπορούμε να ακολουθήσουμε ακριβώς το παράδειγμα της Γερμανίας, θα δεχθώ όχι μόνο φθήνουσα, αλλά αυστηρή αναλογικότητα. Όλοι λέτε ότι είστε φεντεραλιστές, αλλά κανείς δεν θέλει να δεχθεί την αρχή ε, των Ηνωμένων ε, Πολιτειών ε, ή της Γερμανίας, ένα κράτος, μία ψήφος στο δεύτερο σώμα, στο άλλο σώμα, στο έτερο σώμα. Γιατί πάντοτε προσπαθούμε να απομονώσουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από τους υπόλοιπους θεσμούς. Ε, κακώς το κάνουμε αυτό. Δεν είναι αποδεκτό γιατί δεν είναι δίκαιο. Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για όσους ε, είναι πραγματικά υπέρμαρχοι της, ομο... Ομοσπονδίας, αν πιστεύετε ότι όσοι ζουν στο Ζάρλαντ ε, ή στη Βρέμη ε, θεωρούν ότι η σύνθεση της Bundesrat, της Bundesrat είναι ε, δίκαιη, τότε θα μπορούσατε να δεχθείτε τους ίδιους κανόνες ε, στο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο. Μία ψήφος, ένα κράτος. Τότε, αν γινόταν κάτι τέτοιο, θα είχαμε πραγματικά μια δίκαιη σύνθεση και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όταν όμως είμαστε κράτη που έχουν δημογραφικό το κριτήριο στο Συμβούλιο και έχουμε κάτι διαφορετικό στο Κοινοβούλιο, ε, νομίζω ότι είναι σαφή τα πράγματα. Εγώ σέβομαι το, το ότι πιστεύετε ότι στο Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να αλλάξουμε ή ότι δεν θα έχουμε, πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή τότε όμως θα πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη αλλαγή στο Κοινοβούλιο. Για μένα αυτό είναι σαφές. Και θα ήθελα εν τέλει να πω ότι επιμένω, εξακολουθώ να επιμένω ότι έχουμε αυτό το πρόβλημα Αυστρίας και Σουηδίας και ότι πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα. είναι ένα πρόβλημα η κατανομή μεταξύ Αυστρίας, Ουγγαρίας και Σουηδία. Δεν έχω τίποτα απολύτω ε, με την Αυστρία, αντιθέτως, αλλά για τις μεσαίου μεγέθους χώρες που θα χάσουν μία, μία έδρα, νομίζω ότι τουλάχιστον είναι δίκαιο να υπάρχει πλήρης σεβασμός της φθήνουσας ε, ε, αναλογικότητας, ώστε να προσπαθήσουμε να πείσουμε την κοινή μας γνώμη ότι αυτή η συμφωνία αυτή η συνένεση στην οποία ε, καταλήγουμε είναι δίκαιη και ότι ε, είναι ίση για όλους. Καταλαβαίνετε ότι για την Πορτογαλία δεν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον κατά πόσο έχει 20 η Αυστρία και 19 η Σουηδία. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα ε, παθιάσει ιδιαίτερα το, τους ψηφοφόρους μας, αλλά τέλος πάντων είναι σημαντικό να έχουμε έναν κανόνα που θα είναι δίκαιος για όλους. Ναι, αυτό είναι σημαντικό για την κοινή γνώμη και για, την, ε, για να την πείσουμε. Αυτή είναι η μόνη μου παρατήρηση. Εντάξει, δεν είναι ουσιαστική βέβαια. Γιατί θα ήθελα να πω και πάλι, όπως ξεκίνησα άλλωστε, ακόμη και αν είναι δύσκολο για μας να χάνουμε μία ε, έδρα, πρέπει να πω ότι πρέπει να επενέσω την ευρωπαϊκή προσπάθεια που κατέβαλαν ε, οι συνάδελφοί μας και θα ήθελα πραγματικά να τους συγχαρώ για το αποτέλεσμα αυτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είμαι. Δεν θα παρατείνω τη συζήτηση. Οι δύο εισηγητές μας ε, επιχείρησαν εδώ τον τετραγωνισμό του κύκλου. Και πιστεύω ότι συμφωνούμε ότι θα χρειαζόταν μεταρρύθμιση της συνθήκης και αυτό που αποφασίσαμε το 2009 να το συμπληρώσουμε με αλλαγή του εκλογικού νόμου και να ε, ξυγχρονίσουμε την νομοθεσία σχετικά με ευρωπαϊκά κόμματα κλπ. Και να μπορέσουμε να απεικονίσουμε σωστά τα δημογραφικά μας δεδομένα, τα καινούρια. Δεν ε, διαφωνεί κανείς εδώ Οπότε αυτό που πρέπει να σκεφτούμε είναι πώς με την προσχώρηση της Κροατίας θα καταλήξουμε σε μια σωστή αποτύπωση της κατάστασης στην Ευρώπη δημογραφικά. Ε, πρέπει λοιπόν να υπάρχει συμβιβαστική τροπολογία και περιμένω εδώ αν η, ε, θα αντικατοπτρίζεται η προσέλευση στις εκλογές ε, το 2014 σωστά. Και βέβαια οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να δουν ότι η Επιτροπή μας προσπαθεί πραγματικά να ε, βρει μια συμβιβαστική λύση. Και Στι συμβαστικέ ελπίζω να λέει ότι μετά το 2014 θα πρέπει το ταχύτερο δυνατόν να γίνει μια μεταρρύθμιση ριζική σε σχέση με την κατανομή των εδρών. Και θα με ενδιέφερε και ελπίζω μέσα από τις συμβιβαστικέ τροπολογίες που ελπίζω να μας ε, υποβληθούν ε, σύντομα, να μας δείξουν ένα δρόμο εξόδου από το δίλημα και πώς ε, θα μπορέσουμε να κινηθούμε σε σχέση με την αλλαγή της συνθήκης μέσα από συνέλευση ή με άλλο τρόπο. Σίγουρα χρειάζεται πάντο, πάντως μια δημοκρατική διαδικασία και στα κράτη-μέλη που θα λάβει υπόψη της, ε, τα καινούργια δεδομένα ε, της διαδικασίας ολοκλήρωσης. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διαδηλώσουμε την προθυμία μας και να καταστήσουμε σαφή τη θέση μας ότι στα πλαίσια της αναγκαίας επεξεργασίας των συνθήκων και δεν θα ε, γλιτώσουμε την αλλαγή της συνθήκης, να δούμε σε συνολικότερο πλαίσιο το ζήτημα της αντιπροσωπευτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όλα τα νομοθετικά όργανα θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Και υπ' αυτή την έννοια ελπίζω ότι η ε, συμβιβαστική λύση που θα βρούμε θα σημάνει ότι αρχίζει η Επιτροπή μας να μιλάει με μια κοινή γλώσσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Ρέγνερ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Δύο να θα πω. Καταρχήν προς την κατεύθυνση του κυρίου Χέφνερ, να τον στηρίξω δηλαδή και να πω ότι είναι απαραίτητο αμέσως με την επόμενη, στην αρχή της επόμενης θητείας να λύσουμε το πρόβλημα και να μην το αναβάλουμε άλλο. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό δεν μας ε, ωφελεί τώρα, γιατί τώρα πρέπει να λάβουμε μία απόφαση και να βρούμε μία λύση. Πρέπει λοιπόν να συγχαρώ τους δύο εισηγητές που είχαν χάρη καθήκον να εκπληρώσουν και ίσως δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιηθούμε 100% όλοι. Γι' αυτό οι συγητές μας έκαναν το σωστό, δηλαδή ανέπτυξαν βασικές αρχές τις οποίες ετήρησαν. Ε, Ουγγαρία, Σουηδία, Αυστρία, βλέπουμε την αναλογία. Ε, ε εδώ ε, κουτσένει λίγο το πράγμα για να το πω ε, ήπια. Ε, κάποια πράγματα δεν ισχύουν, ιδιαίτερα αν δούμε την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας, αλλά αν το δούμε πιο προσεκτικά το θέμα, εδώ υπάρχει μια δυσαναλογία πρωτίστως λόγω των διαφορετικών πληθυσμών ή μάλλον δεν ταιριάζει στον πληθυσμό Σουηδίας και Ουγγαρίας ή μάλλον λαμβάνεται υπόψη ο πληθυσμό, αλλά όχι οι έδρε. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι έχει πολλέ έδρε η Ουγγαρία. Ε, οι δύο εισηγητέ προσπάθησαν να ε, εφαρμόσουν αυστηρού κανόνε και τον κανόνα ότι δεν μπορεί να χαθεί παραπάνω από μία έδρα και κατέληξαν ότι Ε, αν αλλάζαμε το, τη μέθοδο αυτή, τότε τα αιτήματα θα πολλαπλασιάζονταν. Έτσι λοιπόν η λύση που προτείνουν οι δύο συνεισηγητές είναι σε τελευταία ανάλυση η καλύτερη, η μόνη σωστή. Αλλιώς και επανέρχομαι στην Αυστρία και στην ιδέα να αφαιρεθεί μια έδρα από την Αυστρία. Πρώτον, δεν θα τηρούνταν οι κανόνες και ε, έγιναν, ε, δεν ακούγεται καλά η ομιλήτρια γιατί υπάρχουν παράσιτα. Ε, θα λύναμε, ε, έτσι πρέπει να προσέξουμε η αδικία που τώρα αφορά τη Σουηδία να μην μεταφερθεί στην Αυστρία. Τώρα μπορούμε να βρούμε κάποια λύση ρεαλιστική που να είναι και λογική. Να δούμε τώρα ποιος θα ζητεί το λόγο. Ο επόμενος. Δεν ζητεί κανείς το λόγο. Οπότε ξαναγυρίζουμε στους ε, συνεισηγητές για να απαντήσουν. Chairman, I, I, Δεν χρησιμοποίησα το δικαίωμα του λόγου που είχα μέχρι τώρα, γιατί συμφώνησε καταρχήν με τον κύριο Φόξ ότι δηλαδή εάν πάρουμε την έδρα από την Ουγγαρία αυτό δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι υπάρχει αδικίες βάρος της Σουηδίας. Νομίζω ότι κύριε Φο... η κυρία που μίλησε πριν ε, είπε κάτι που δεν είναι ακριβές, μήπως θέλετε να με διορθώσετε. Ευχαριστώ. Αυτό που είπα εγώ είναι το εξή. Αν δείτε τον πληθυσμό Ουγγαρίας και Σουηδίας, υπάρχει διαφορά περίπου 500.000 άνθρωποι. Η Ουγγαρία και η Σουηδία είναι κοντά σε σχέση με τον πληθυσμό που έχουν. Τώρα η Ουγγαρία έχει 22 έδρες και η Σουηδία 20, παρόλο που δεν είναι μεγάλη η πληθυσμιακή τους διαφορά. Η σχέση μεταξύ Σουηδίας-Αυστρίας έχει ως εξής. Υπάρχει διαφορά περίπου ενός εκατομμυρίου. Δηλαδή στη Σουηδία ο πληθυσμός είναι μεγαλύτερος κατά ένα ε, εκατομμύριο και έχουμε 20 με 19 διαφορά ψήφων. Τώρα, ε, τι προτείνουν οι συγητές. Να χάσει η Ουγγαρία μία έδρα και να χάσει και η Σουηδία και τότε πράγματι η σχέση Αυστρίας-Σουηδίας είναι σχετικά ισορροπημένη, αλλά η σχέση Ουγγαρίας-Σουηδίας δεν αλλάζει πολύ. Υπάρχουν πάλι, υπάρχει πάλι μια διαφορά δύο εδρών. Υπ' αυτή την έννοια η δικαιότερη λύση θα ήταν να χάσει δύο έδρες η Ουγγαρία σύμφωνα και με την αρχή της φθήνουσας αναλογικότητας, αλλά αυτό πάλι αντιφάσκει προς τις βασικές αρχές που προτείνουν οι δύο μας εισηγητές. Αυτό που εννοούσα εγώ είναι ότι η σχέση Σουηδία-Αυστρία μετά θα είναι μια άδικη σχέση. Θα είναι το πρόβλημα που υπάρχει τώρα ας πούμε μεταξύ Ουγγαρίας και Σουηδίας το οποίο μετατοπίζεται ως άδικη σχέση μεταξύ Σουηδίας και Αυστρίας. Δεν θα ήταν τόσο ακραίο όπως είναι στη δυσαναλογία Ουγγαρία-Σουηδία παρόλα αυτά όμως θα υπήρχε μια σχετική αδικία και εις επίμετρον υπάρχει και αντίφαση προς τις βασικές αρχές τότε που έθεσαν δύο εισηγητές. Ο κύριος Γκουαλτιέρη, ο κύριος Τσασκόφσκι να απαντήσουν παρακαλώ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα σας τα σχόλια. Όσον αφορά τις συμβιβαστικέ τροπολογίες, ε, τις ε, οριστικοποιήσαμε πριν από δύο ώρες. Κανονικά η γραμματεία θα έπρεπε να σας τις υποβάλει πριν από την συνεδρίαση. Συγγνώμη αν δεν έγινε αυτό και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δύο σχόλια έχω βασικά. Πρώτον, όσον αφορά το ερώτημα, το θέμα Σουηδία-Αυστρία. Το συζητήσαμε πολλές, πολλές φορές και το εξηγήσαμε. Αν θέλουμε να έχουμε αν θέλουμε να έχουμε τη σωστή αναλογία πληθυσμού ε, εδρών, πρέπει από κάποια κράτη-μέλη να αφαιρέσουμε πάνω από μία έδρες και είδαμε, δείξαμε το, το, την προσέγγιση μας, στάδιο 1, 2, 3 κλπ. Και παρουσιάσαμε το συλλογισμό μας. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στο παρελθόν είχαμε ομάδες χωρών και έτσι φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα. Αν δει κανείς όμως τον τελευταίο πίνακα και αν δει για παράδειγμα την αναλογία πληθυσμού και εδρών, ε, μπορεί κανείς να υποκαταστήσει τη Σουηδία με την Αυστρία. Δεν θελήσαμε να αλλάξουμε τα νούμερα γιατί δεν θελήσαμε να ε, αμφισβητήσουμε τη λογική πίσω από αυτά. Όμως πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την τροπολογία που έχει υποβληθεί γιατί από ό,τι βλέπω έχει την υποστήριξη μεταξύ κάποιων συναδέλφων μας ε, και επίσης από την ε, πολιτική μου ομάδα υποστηρίζεται. Γιατί υπάρχει μια λογική αν περνάει κανείς από διάφορα στάδια και αν έχει κανείς ομάδες χωρών και είναι και μια άλλη λογική όταν βλέπει κανείς μόνο τον τελευταίο πίνακα και ορισμένοι άνθρωποι θα κοιτάξουν μόνο τον τελευταίο πίνακα. Οπότε Πιστεύω ότι αυτό είναι που πρέπει να αποφασίσει πρώτα η Επιτροπή μας μέσω ψηφοφορίας και μετά η Ολομέλεια όσον αφορά τώρα το μαθηματικό τύπο όλοι συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα, μια μόνιμη διαφανής λύση στο πρόβλημα και συμφωνούμε ότι μπορούμε να το επιτύχουμε αυτό μόνο όταν υπάρχουν ε, και τα άλλα θεσμικά παζλ ε, στο τραπέζι. Αν είναι να αποφασίσουμε από τώρα για το μέλλον, τι είδου τύπο, κατά πόσο θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε καν μαθηματικό τύπο και τι είδου τύπο θα έπρεπε να είναι αυτός, ε, νομίζω ότι δεν θα φτάσουμε σε συνένεση. Υπενθυμίζω στους συναδέλφους ότι εγώ ήμουν το μόνο μέλος της Επιτροπής μας, εκτός από, τον οργάνω, από την οργάνωση ε, της ε, ε, διάσκεψης στο Cambridge, ήταν εκεί και ο Άντριου Νταφ, ε, το θέμα είναι το εξή όμως. Αν πρέπει να αποφασίσουμε ότι θα γίνει επί της βάσης μαθηματικού τύπου, μπορούμε να αποφασίσουμε επ' αυτού μόνο αν αποφασίσουμε και άλλα θεσμικά θέματα. Αν θέλουμε να πούμε είναι μαθηματικός ο τύπος και ότι πρέπει να είναι αυτός ο μαθηματικός τύπος και όχι κάποιος άλλος, τότε δεν θα υπάρχει συνένεση. Άρα, ανεξαρτήτως των δικών μου προσωπικών ε, απόψεων επ' αυτού. Γι' αυτό ακριβώς δεν το συμπεριλάβαμε στο κείμενο και δεν σημαίνει ότι δεν συμφωνούμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μια μόνιμη λύση και ότι θα ήταν αυτό καλύτερο από το να ε, τα εξετάζουμε κάθε τρεις και λίγο. Όμως αυτή τη στιγμή για την ώρα αυτό το θέμα δεν τίθεται. Γι' αυτό δεν το συμπεριλάβαμε σε καμία από τις συμβαστικές μας λύσεις. Όταν όμως ασχοληθούμε με το ζήτημα αυτό στο μέλλον ε, και ε, μάλλον κάποιος άλλος θα το κάνει. Ε, ελπίζω κάποιος άλλος να το κάνει. Ε, θα ε, βρούμε μία λύση που θα την ξανασυζητήσουμε πολλές φορές. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω οι συμβιβαστικές τροπολογίες που προετοιμάσαμε να είναι μία καλή λύση συμβιβασμού με τους σκιώδεις εισηγητές, με τους οποίους θα συνεδριάσουμε μετά το τέλος της σημερινής μας συνεδρίασης. Για να... Έχετε κάτι να προσθέσετε, κύριε ναι, για να ενημερώσω τους συναδέλφους. Πού έχουμε κάνει την συνάντηση και δοσηγητές για να συζητήσουμε αυτή την συμβαστική πρόταση που ακόμα δεν έχουμε στείλει στη γραμματεία και πρόκειται για αυτό το οποίο Σα έχουμε εξηγήσει, οπότε και εγώ πιστεύω ότι βάσει τη συζήτηση που έγινε ότι έχουμε δεδομένες τι προποθέσει για να έχουμε ένα ευρύτατο μια ευρύτατη συνένεση για αυτόν τον συμβασμό, οπότε και έτσι θα στείλουμε και ένα ισχυρό πολιτικό μήνυμα. Οπότε από μια μεριά να γνωρίζει το Κοινοβούλιο την αναγκαιότητα του θα πρέπει να υπάρχει ένας αντικειμενικός μηχανισμός. Και επίσης δεσμευόμαστε να αναλάβουμε κάποια πρωτοβουλία τέλος πάντων και από την ελληνική όπω όπως είπε ο συνάδελφος ε, να γνωρίζετε ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν εκτός του πλαισίου κάποιες γενικότερες αναθεώρησης και προβληματισμού τέλος πάντων τουλάχιστον όσον αφορά την ισορροπία μεταξύ των δύο μηχανισμών των δύο θεσμικών οργάνων Συμβουλίου και Κοινοβουλίου γιατί ακριβώς ορίζουν οι συνθήκες ότι είναι το θεμέλιο της Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας η αντιπροσώπευση των πολιτών και των κρατών μελών. Επίσης είναι σαφές ότι πάρα πολύ δύσκολα μπορούμε να προχωρήσουμε προς ένα ακραίο πρότυπο και να έχουμε ε, σε ένα κοινοβούλιο τους πολίτες και σε άλλο δηλαδή, τα κράτη-μέλη, έχουμε μεικτό σύστημα για προφανείς λόγους. Πάντως από την άλλη μεριά είναι σωστό ότι με αυτόν τον τρόπο που γίνεται η κατανομή αυτού του, του, του, μείγματος ε, προσώπων ε, και κρατών μελών στο Κοινοβούλιο, αυτό ε, μπορεί να ρυθμιστεί πολλούς τρόπους, οπότε και γι' αυτό είναι ξεκάθαρο ότι αν γίνει η αλλαγή που αφορά τα, τα πρόσωπα θα γίνει η αλλαγή και όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιηθούν και τα δύο κριτήρια να συντρέχουν και για τη σύνθεση του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου. Επομένως έχουμε εδώ στην συνθήκη μία συμμετρία όσον αφορά το, το ότι ξεκάθαρα με ακρίβεια ορίζεται τι ισχύει για το Συμβούλιο αλλά όχι για αυτή την ε, φθήνουσα αντιπροσωπευτικότητα. Γιατί είπαμε ότι μπορούμε να έχουμε μαθηματικό τύπο που να στηρίζει τη ρύθμιση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε μια συνένεση, σε μια δέσμευση και στο δυνάμει αναθεώρηση της συνθήκης όσον αφορά τους αριθμούς, τα αριθμητικά στοιχεία για τη Σουηδία, την Αυστρία. Εδώ έχουμε ένα συγκεκριμένο θέμα. Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε κάποιες ε, κάποιες, κάποιες τροποποιήσεις, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε πει να απορριφθεί... Τέλο πάντων υπάρχουν επιχειρήματα και προς τις δύο κατεύθυνσεις για το συν και για το πλήν. Έχουμε προτίμηση, αλλά καταλαβαίνουμε για την αντίθετη λογική και θα μπορούσε κάποιο τρόπο έτσι να γίνει αυτή η θυσία ως πως ε, αυτές τις δύο χώρες, Σουηδία και Αυστρία, δεν θέλαμε να γίνει κάποια πιο απλή ε, κατανομή των εδρών και επίσης να έχουμε αυτή τη διαφορά των δύο εδρών μεταξύ Ουγγαρίας και Σουηδίας. Αυτό προϋπήρχε, δεν το εφήβραμε εμείς, αλλά γι' αυτό και το Κοινοβούλιο αποφάσισε με πολύ ευρεία συνένεση να γίνει αυτή η κατανομή και έτσι είχαμε αυτή την διαφορά των δύο ευρώ. Δεν είναι υποχρεωτικό, θα μπορούσαμε να πούμε τρεις, τέσσερις, παραπάνω Σουηδία, να πάνε κάπου αλλού. Οπότε... Αυτό είναι το θέμα που επισημάνθηκε. Επισημάνθηκε ότι δίνει μια χρειά άδικη στην πρότασή μας. Αλλά προϋπήρχε αυτή η διαφορά. Το πιο λογικό θα ήταν, όπως είπαμε στην πρώτη φάση, να πάρουμε μια έδρα από την Ουγγαρία, αλλά να μην το κάνουμε αυτό. Ακριβώς λόγω της αρχής του να μην χάσει, να μην κερδίσει κανείς πάνω από μία έδρα. Επομένω, υπάρχει μια συγκεκριμένη λογική στην πρότασή μας από την άλλη μεριά, όμως θα μπορούσε κανείς να πει τα ίδια και για τα αντεπιχειρήματα. Γι' αυτό σας λέω, για μας αυτό δεν είναι κόκκινη γραμμή. Να δούμε τι θα πρεσβεύει η πλειοψηφία στην Επιτροπή. Και ό,τι αποτέλεσμα και να βγει, είμαι βέβαιος ότι όσο είναι δυνατόν, μπορεί να μην είναι η πρότασή μας τέλεια, αλλά είναι ρεαλιστική, βιώσιμη. Και γι' αυτό και επιθέλουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ευρεία στο Κοινοβούλιο. Αν και αν συμβεί κάτι τέτοιο, τότε ίσως το Συμβούλιο συμφωνήσει. Γιατί θα γίνουν εκλογές και θα έχουμε και την προσχώρηση της Κροατίας. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Νταφ. Έχετε το λόγο. Για ένα σημαντικό θέμα θα ήθελα να μιλήσω. Ο Ρομπέρτο λέει ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε την τρέχουσα σύνθεση του Κοινοβουλίου. Όχι. δεν έγινε κάτι τέτοιο. Αντιθέτως ήταν τμήμα ε, του συμβιβασμού για τη Λισαβόνα η τρέχουσα σύνθεση και εμείς δεν, ε, είχαμε, δεν είπαμε καθόλου την άποψή μας ε, ως προς αυτό. Και επειδή εγώ ήμουν ένας από τους διαπραγματευτές που ένας από αυτούς που συμμετείχε ε, στους, στις διαπραγματεύσεις μαζί με τον Μπαρόν Κρέσπο και τον ε, ε, Μπροκ. Εμείς διαφωνούσαμε με, διαφωνήσαμε με την, με, με την τρέχουσα σύνθεση Πιστεύω ότι με τη σοφία της Επιτροπής μας αλλά και των συνεισυχητών θα επιτύχουμε αυτή τη φορά ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Και πραγματικά έχω αρχίσει να στεναχωριέμαι που η Αυστρογγαρία διαλύθηκε, γιατί αυτό θα μας είχε λύσει το πρόβλημα, να σας πω την αλήθεια. Uh, Μία σύντομη απάντηση, κύριε Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως δεν ναι, ενέκρινε ναι, τη σύνθεση, τη, τη σύνθεση αυτή ε, ε, γιατί δεν υπήρχε φυσικά τότε η συνθήκη της Λισαβόνας και δεν είχαμε αυτή τη διαδικασία. Όμως, ε, βάσει άλλου συνολικού αριθμού, 750, ενέκρινε την έκθεση Σεβερίν Λαμασούρ που πρότεινε την προσθήκη ε, κάποιων εδρών σε κάποια κράτη-μέλη, κάτι το οποίο οδήγησε στη διαφορά ε, δύο εδρών μεταξύ ε, Ουγγαρίας και Σουηδίας. Το προηγούμενο κοινοβούλιο το είχε υπερψηφίσει αυτό. Αυτό εννοώ. Δεν είπα ότι ενέκρινε την θέση μέσω της σύμφωνης γνώμης, γιατί αυτό είναι μια διαφορετική διαδικασία, αλλά τέλος πάντων αυτή η ψηφοφορία έλαβε χώρα. Point of I mean διαδικαστικά. Κρίνοντας από το οικογενειακό μου ιστορικό, εγώ θα ήμουν υπήκος της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας, οπότε διαφωνώ κάθετα. Θέλω πολλά προβλήματα και επομένω. Αύριο θα συνδυάσουμε 10 με 3. Αλλά δεν ξέρω. Ίσως οι σκιώδες ηγητές και οι ηγητές μπορούν να παραμείνουν και οι διερμηνείς μέσα σε 7 η ώρα. Τους υπόλοιπους θα σας δω αύριο. 9 η ώρα αύριο οι συντονιστές μου το ξεχνάτε.